Μπορούμε να αρχίσουμε. Καλημέρα σε όλους. Σας, θυμ... Σας θυμίζω ότι αναμεταδίδεται η συνεδρίασή μας μέσω του διαδικτύου. Η ημερήσια διάταξη 28 Σεπτεμβρίου του 2011 μοιράστηκε. Και αν δεν έχετε αντιρρήσεις εγκρίνεται. Ανακοινώσεις Πρόεδρου. Θυμίζω ότι στη συνεδρίαση της 28 Σεπτεμβρίου οι συντονιστές συμφώνησαν για ορισμένους διορισμούς, τις οποίες, τους οποίους θα σας διαβάσω και αν δεν έχετε παρατηρήσεις εγκρίνονται. Διαδικασία διαβούλευσης ε, και ε, σχετικά με τις εγγυήσεις για την Ιρλανδία. Θέλησε η Ιρλανδία η δήλωση ε, να, μεταβληθεί σε πρωτόκολλο. Και κανένας δεν έφερε αντιρρήσεις, ο Ίνιγκο είχε μια επιφύλαξη, δεν ξέρω αν μπορεί να την άρει. Τώρα, για τις επιλογές για την Τσεχία το ίδιο πράγμα πρόκειται για την ε, για τη δήλωση παράρτημα στη συνθήκη της Λισαβόνας που πρέπει να γίνει πρωτόκολλο. Και η συγητής θα είναι ο κύριος Νταφ. Τι τρέχει, αλήθεια λέει ο πρόεδρος. Γνώμοδότηση για την άφετε σχετικά με την προσχώρηση της Κροατίας. Οι συντονιστές διόρισαν τον κύριο Τρασκόφσκι Γνωμοδότηση για την ε, ΛΥΜΠΕ σχετικά με το έτος της ε, Ιθαγένειας του 2003. Ο κύριος Χέφνερ από τους Πράσινους έχει την εισήγηση. Και ο κύριος Δάφ και πάλι θα είναι εισηγητής ε, για την τροποποίηση του κανονισμού σχετικά με τις ψηφοφορίες με ονομαστική ψηφοφορία στις επιτροπής. Υπάρχει πρόταση η τελική ψηφοφορία να γίνεται πάντα στις επιτροπές ηλεκτρονικά. Και αν κανείς δεν έχει παρατηρήσεις, ούτω συμφωνείτε. Εγώ θα στείλω μία επιστολή στον κύριο Μπαρόσο για να τον πληροφορήσω ότι στις επόμενες συνεδρι... να έρθει σε μία από τις επόμενες συνεδριάσεις για να συζητήσουμε για τις προοπτικές με τροποποίησης των συνθήκων για την οικονομική governance. Και αν κάτι τέτοιο φυσικά ε, συμβεί, δηλαδή αν η υπόθεση ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα διατυπώσει προτάσεις, τότε θα καλέσουμε φυσικά τον κύριο Βαν Έγκριση των πρακτικών των προηγουμένων συνεδριάσεων. Είναι στη διάθεσή σας ενιαίο πρακτικό της 7ης Σεπτεμβρίου του 2011. Αν δεν μου έχετε στείλει παρατηρήσεις, τώρα δεν πρόκειται να δεχθώ καμία, οπότε το εγκρίνω. Πάμε τώρα στο πιο σημαντικό σημείο της συνεδρίασής μας σήμερα. Αφορά στη στροποποίηση στον κανονισμό για τον κώδικα συμπεριφοράς στο Ευρωκοινοβούλιο σχετικά με τα οικονομικά συμφέροντα και το ασυμβίβαστο Λοιπόν, έχουμε τον κώδικα συμπεριφοράς ε, που θα συνταχθεί από την ομάδα που συντάχθηκε από την ομάδα εργασίας και μετά πρέπει να περάσει από τη διάσκεψη των Προέδρων. Συζητήθηκε, παρουσιάστηκε το κείμενο, δεν έχω παρατηρήσει, δεν έλαβα ιδιαίτερες παρατηρήσεις, Συζητήσει είμαι εγώ. Και εγώ παρουσιάζω την έκθεσή μου λέγοντας και θυμίζοντας ότι αρμοδιότητες αυτής της Επιτροπής ε, είναι η τροποποίηση του κανονισμού βάσει του άρθρου 232 της Συνθήκης. Εμείς είμαστε δηλαδή που πρέπει να τροποποιήσουμε αυτόν τον κανονισμό. Σημαίνει λοιπόν ότι αυτός ο κώδικας συμπεριφοράς θα πρέπει να ενσωματωθεί μέσα στον κανονισμό. Εγώ παρουσιάζω το κείμενο έτσι όπως βγήκε από την ομάδα εργασίας και τη διάσκεψη των Προέδρων. Και ουσιαστικά Θέλω να προχωρήσουμε γρήγορα χωρίς να τροποποιήσουμε ιδιαίτερα το κείμενο. Υπάρχει βέβαια μεταξύ των άλλων κάποιο προβληματάκι και το ανέφερα την προηγούμενη φορά. Δεν θέλω να ξαναπώ, να, αναφέρω εδώ και πάλι το κείμενο, διότι θα έχανα χρόνο. Να σας θυμίσω, προβλέπει γενικές αρχές συμπεριφοράς, προβλέπει την υποχρέωση δήλωσης ε, για τα οικονομικά συμφέροντα στην αρχή της κοινοβουλευτικής θητείας προβλέπει κυρώσεις σε περιπτώσεις παραβίασης του κώδικα συμπεριφοράς και προβλέπει κυρίως ε, ε, κανόνες, σαφείς κανόνες που υπολογι... με αριθμητικά ονομαστικά ποσά σε ευρώ για σχετικά με δώρα κλπ. Ο κανονισμός ήδη προβλέπει το άρθρο 19, είναι αλήθεια. Ναι, ναι, το 19, το 19. Το 9, το 9, α, το 9 είναι λόρ, τότε. Ε, προβλέπει το άρθρο 9 που αναφέρεται στον προηγούμενο κώδικα συμπεριφοράς. Και το πιο λεπτό θέμα είναι το θέμα των κυρώσεων, των ποινών. Διότι η ομάδα εργασίας, το έγγραφο της ομάδας εργασίας αναφέρει έναν αριθμό κυρώσεων που είναι οι ίδιες με το εκείνες του άρθρου 153 του κανονισμού εκτός από μία ποινή, μία κύρωση παραπάνω και εδώ θα πρέπει να με βοηθήσετε με τη συμβουλή σας. Οι κυρώσεις του 153 εντάσσονται μέσα στο πλαίσιο της εσωτερικής πειθαρχίας Είναι γενικού χαρακτήρα λοιπόν κυρώσεις. Ο κώδικας συμπεριφοράς που σας επιβάλλω αναφέρει όλες αυτές τις κυρώσεις χωριστά στο εσωτερικό του κώδικα συμπεριφορά που θα γίνει παράρτημα 1. Τώρα για λόγους ε, νομοθετικής απλούστευσης που πάντοτε μας τη ζήτησαν να αφαιρέσουμε το άρθρο 153 δεδομένου ότι αφορά τις ίδιες κυρώσεις. Αυτή είναι η γνώμη μου. Καλό θα ήταν ε, να αφήσουμε μόνο τον κώδικα συμπεριφοράς. Εγώ πιστεύω ότι για νομοθετική απλούστευση να αφαιρέσουμε το άρθρο 153. Προστίθεται όμως μία κύρωση. Ανάκληση της ε, εντολής ως εισηγητού ενός βουλευτή. Πρόκειται για κάτι το πολύ λογικό, πρόκειται για κάτι το νέο, μιλάμε για διαφάνεια της κοινοβουλευτικής εργασίας. Ο εισηγητής μπορεί κάλλιστα να υποστεί πιέσεις, άρα μπορούμε, ε, ε, είναι λογικό να τον ανακαλούμε. και πώς εμείς ε, να εισάγουμε, να τακτοποιήσουμε αυτή την κύρωση άμα κρατήσουμε το άρθρο 153 θα πρέπει να προσθέσουμε αυτή την ποινή και στο άρθρο 153 και υπάρχει και κάτι άλλο ουσιαστικό οι εφαρμοστικές λεπτομέρειες ορίζονται των κυρώσεων ορίζονται στο άρθρο 19. Και το άρθρο 19 προβλέπει ότι ο πρόεδρος είναι αυτός που είναι αρμόδιος για την εφαρμογή των κυρώσεων. Αλλά για την ανάκληση μιας εκλογικής εντολής, ενός εκλογικού αξιώματος, δηλαδή πρόεδρος, αντιπρόεδρος, πρόεδρος επιτροπής κτλ. Για αυτό προβλέπεται με μια ειδική πλειοψηφία ε, να το κάνει η διάσκεψη των Προέδρων και μετά να το υποβάλει στην Ολομέλεια. Μπορούμε το ίδιο σύστημα να το εφαρμόσουμε και στην ανάκληση της εντολής ως εισηγητή. Η ομάδα εργασίας λέει για την ε, κύρωση που αφορά στην ανάκληση του εκλογικού αξιώματος περιορίζεται να και λέει προτείνεται η κύρωση στη διάσκεψη των πρόεδρων αλλά δεν, το, δεν επαναλαμβάνει το ίδιο με αυτό που σας ανέφερα προηγουμένως για την ανάκληση δηλαδή του εκλογικού αξιώματος. Προτείνω λοιπόν εγώ στην έκθεσή μου να θεωρήσουμε τον διορισμό ως εισηγητή αντίστοιχα με το, την εκλογική εντολή. Οπότε για την ανάκληση του διορισμού ως εισηγητή να χρησιμοποιήσουμε την ίδια διαδικασία με εκείνη της ανάκλησης των κοινοβουλευτικών αξιωμάτων. Λοιπόν, λέει ότι ένα από τα αξιώματα είναι και η ανάθεση εισήγηση. για την ανάκληση του αξιώματος του εισηγητή προστρέχουμε στο άρθρο 153, στις διαδικασίες που προβλέπει το άρθρο 153. Ποια είναι η δυσκολία τώρα και, σας, και θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας. Θα μπορούσα βέβαια να καταθέσω και μία τροπολογία αν δεχτείτε αυτήν τη δεύτερη υπόθεση που εγώ σας προτείνω. Το πρώτο λοιπόν που τίθεται είναι το εξή. Αν θεωρήσουμε το αξίωμα του εισηγητού ως εκλογικό αξίωμα ε, είναι πραγματικά κάτι το τραβηγμένο. διότι αναθέτουμε μία εισήγηση μετά από συζήτηση μέσα στους συντονιστές και αξιοποιούμε πόντους που έχουν στη διάθεσή τους οι ομάδες. Αυτό είναι το καθαρά τυπικό και το ξεπερνάμε. Υπάρχει κατά τη γνώμη μου όμως κάτι πολύ πιο ουσιαστικό. Είναι η αναλογικότητα των κυρώσεων. Έχουμε την πιο βαριά κύρωση που είναι η ανάκληση του αξιώματος. Τώρα, εδώ, επειδή είναι πολύ σοβαρή η ποινή, ε, θέλουμε να δώσουμε εγγύηση στην όλη διαδικασία. Αλλά δεν είναι ένας πρόεδρος ο οποίος ανακαλεί, αλλά είναι η διάσκεψη των πρόεδρων και μετά η Ολομέλεια. Μπορούμε να κάνουμε το ίδιο πράγμα και για το αξίωμα του εισηγητή. Σίγουρα στο θέμα της ανάθεσης μια συζήτηση εισήγησης έχουμε σημαντικές πολιτικές αρμοδιότητες αλλά δεν είναι το ίδιο με την ανάκληση να σε ανακαλούν από αντιπρόεδρο, πρόεδρο επιτροπής ή κοσμήτωρα κτλ. για την ανάκληση των στρίκτου ένσου εκλογικών αξιωμάτων είναι λογικό να αποφασίζει η Ολομέλεια, διότι η Ολομέλεια είναι αυτή που αναθέτει το αξίωμα. Αλλά για τον εισηγητή, ε, το αξίωμα του εισηγητή το δίνει η αρμόδια επιτροπή. Θα μπορούσαμε λοιπόν εμείς να φανταστούμε μία τροπολογία στο κείμενο η οποία θα ανέθετε την αρμοδιότητα ανάκλησης του, διορισμού σε, ε, σε εισηγητή στην αρμόδια επιτροπή. Θέλω να μην πειράξω ιδιαίτερα το κείμενο, αλλά μερικές αλλαγές τυπικού χαρακτήρα πρέπει να γίνουν, εάν θέλουμε δηλαδή εμείς να εκπληρώσουμε τα καθήκοντά μας, δηλαδή να συμπληρώσουμε τον κανονισμό. Υπάρχει βέβαια και η άλλη αλλαγή για την οποία δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν πιστεύω ότι στον τωρινό κώδικα συμπεριφοράς προβλέπεται ότι θα πρέπει να δίνουμε πληροφορίες και για τη συμμετοχή στα intergroup. Αυτό δεν αναφέρεται. Αυτό όμως μου φαίνεται να είναι απλώς ε, ε, απλώς να ξεχάστηκε. Μέσα στο άρθρο 39 βρίσκεται. Το 39, α όχι δεν είναι το 39, το 32 το 32. Ξεκινάμε λοιπόν τη συζήτηση. Γερέρο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Στην αρχή της παρέμβασής σας αναφερθήκατε στη σημασία που επέχει το θέμα αυτό το οποίο συζητάμε σήμερα. Η σημασία αυτή προέρχεται από ένα πολιτικό σενάριο το οποίο αντιμετωπίζουμε μέσα σε αυτή την χρηματοοικονομική και κοινωνική κρίση που οδηγεί και σε μια πολιτική υποβάθμιση και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε πολλές από τις χώρες μας. Βρίσκεται σε δυσκολία ο πολιτικός κόσμος. Κάθε φορά όλο και περισσότεροι πολίτες απορρίπτουν την πολιτική δράση. Άλλοι πολίτες υποστηρίζουν την πολιτική αλλά θέλουν να ασκηθεί με διαφορετικό τρόπο. Αυτό είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε συνέχεια στις δημοσκοπήσεις της ε, χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι εμείς ως πολίτες είμαστε μία από τις μεγαλύτερες πηγές ανησυχίας για τους πολίτες. Επομένως, νομίζω ότι ό,τι μπορούμε να κάνουμε για να αυξήσουμε την νομιμοποίηση της πολιτικής, να αυξήσουμε την διαφάνεια στον πολιτικό χώρο, να υπάρξει μια αναβάθμιση του ρόλου των πολιτικών οργάνων, αυτό είναι θετικό και είναι ακόμα και απαραίτητο. Επίσης, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπουμε να αναδύεται μια κριτική στάση εναντί των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά σημαίνουν <clears throat> ότι για μένα το θεμελιώδες στοιχείο αυτής της έκθεσης που συζητάμε σήμερα να μπορέσουμε να μεταφέρουμε στους πολίτες μας την ιδέα ότι τα θεσμικά μας όργανα είναι διάφανα, ότι οι εκπρόσωποι μας είναι, είναι άτομα τα οποία υπόκεινται σε ένα ηθικό κώδικα, ένα κώδικα συμπεριφοράς, αυτό είναι κάτι το οποίο θα αυξήσει την εμπιστοσύνη σε εμά των πολιτών. Προ την κατεύθυνση αυτή λοιπόν νομίζω ότι το έργο το οποίο είχε φέρει σε πέραση η ομάδα εργασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Προεδρείου μάλλον, είναι μια θετική εργασία και η υποδοχή αυτού του έργου από τον πρόεδρο Κασίνη τη έκθεση αυτή είναι και αυτή πάρα πολύ θετική. Όπω είπε και ο πρόεδρο Κασίνη, Πρόκειται για να μπορέσουμε το ταχύτερο δυνατό να θέσουμε σε εφαρμογή αυτές τις νέες διατάξεις και πρόνοιες που, αυξάνουν την εμπιστοσύνη των πολιτών και τη διαφάνεια του οργάνου μας. Βέβαια έχουμε ξεκινήσει αυτή τη ε, διαδρομή στην ίδια την Επιτροπή μας όταν εγκρίναμε την ε, αναθεώρηση του κατάστοιχου διαφάνειας για τις ομάδες πίεσης, τα λόμπι, και βρισκόμαστε στην ίδια κατεύθυνση, να είμαστε πιο ανοιχτοί προς τους πολίτες, να εξηγήσουμε στους πολίτες τι κάνουμε και να μπορούν οι πολίτες να ελέγχουν καλύτερα τη δραστηριότητά μας, τη συμπεριφορά μας και το καθαρό της πολιτικής μας δράσης. Την καθαρότητα της πολιτικής μας δράσης. Ένα δεύτερο όμως σημείο στο οποίο θέλω να αναφερθώ είναι το θέμα της απλοποίησης, της απλότητος. Η εμπειρία σε πάρα πολλές από τις χώρες μας καταδεικνύει ότι όσο απλούστερη και πιο ευανάγνωστοι και πιο εύκολοι στην εφαρμογή είναι οι κανόνες, τόσο το καλύτερο. Όταν είναι πολύπλοκοι κανόνες που είναι ανοιχτοί σε διάφορες ερμηνείες και που στο τέλος ανήκουν πάντα παραθυράκια για να μπορεί κανείς να αποφύγει την εφαρμογή τους, αυτοί είναι προβληματικοί οι κανόνες. Γι' αυτό εγώ υποστηρίζω την απλότητα, την αμεσότητα <clears throat> των διατάξεων που θα πρέπει να εγγραφούν μέσα σε αυτή τη μεταρρύθμιση που θέλουμε να εφαρμόσουμε. Θεωρώ επίσης θετικό το ότι υπάρχει μια συμβουλευτική επιτροπή η οποία μπορεί να βοηθήσει τους κοινοβουλευτικούς να έχουν σαφήνεια στο μυαλό τους σε σχέση με τις υποχρεώσεις τους και σε σχέση με τα όρια της συμπεριφοράς τους. Συχνά ή τουλάχιστον κάποιες φορές όταν παραβιάζονται κάποιοι κανόνες συμπεριφοράς δεν γίνεται πάντα αυτό με κακή πρόθεση δεν γίνεται ηθελημένα, πολλές φορές γίνεται μόνο λόγω άγνοιας των κανόνων και των ορίων που πρέπει να διέπουν την κοινοβουλευτική συμπεριφορά. Άλλες φορές όμως δυστυχώς δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ο κύριος Σταφ θυμάται σίγουρα, αυτό είναι κάτι το οποίο εγώ το έμαθα όταν ήμουν ακόμα πιτσιρίκος, όταν μπήκα στον δημόσιο μηχανισμό της Ισπανίας, στην δημόσια δίκηση Υπάρχει ένας βρετανικός τρόπος για να αναφέρεται κανείς στους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα και έλεγε ο κύριος Δάφ ότι όταν επιλέγουμε τους ε, δημόσιους υπαλλήλους είναι να είναι έντιμα άτομα. Γιατί αν δεν είναι έντιμα, όσο πιο ικανή είναι, τόσο χειρότεροι θα αποδειχθούν στο μέλλον. Επομένως, το ουσιαστικό στοιχείο εδώ είναι να έχουμε και αυτή τη Συμβουλευτική Επιτροπή η οποία θα είναι σε θέση να διευκρινίσει ακριβώς ποια είναι τα όρια σε κάθε περίπτωση. Επομένως, συνολικά υποστηρίζουμε απόλυτα τις τροποποιήσεις που προτείνει ο Πρόεδρος. Τώρα, σε σχέση με τα προβλήματα που υποδείξατε σε σχέση με το καθεστώς κυρώσεων, εγώ δεν μπορώ τώρα να σας δώσω μια άμεση απάντηση, αλλά η ομάδα μου θα μπορέσει Ελπίζω το ταχύτερο δυνατό να σα δώσω μια απάντηση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή στη γραμματεία της Επιτροπής μας. Αυτό το οποίο θα ήθελα να αναφέρω όμω είναι το εξής. Νομίζω ότι πρέπει να κάνω μια σαφή διάκριση μεταξύ της, ε, ενός ερετού αξιώματος αφενός και του αξιώματος ενός εισηγητή. Η, τα αιρετά αξιώματα έλκονται από του πολίτες. Οι πολίτες είναι αυτοί που έχουν εκλέξει κάποιον βουλευτή και οι λόγοι για τους οποίους πρέπει να υπάρξει ανάκληση μιας τέτοιας ερετής ενός ερετού αξιώματος είναι έκτακτη λόγοι. Στη χώρα μου παραδείγματος χάρη χρειάζεται. Υπήρξε και μια απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Ισπανίας που λέει ότι μόνο για λόγους ποινική καταδίκης που αφαιρεί τα δικαιώματα του βουλευτή ή του γερουσιαστή μπορεί να ανακληθεί η κοινοβουλευτική του εντολή. Επομένως, θα μπορούσαμε ίσως να εξετάσουμε τη δυνατότητα να υπάρχει παράλληλη διαδικασία, να υπάρχει το ίδιο όργανο το οποίο λαμβάνει αποφάσεις και στις δύο περιπτώσεις, αλλά κάνοντας από την αρχή μια σαφή διάκριση ότι η ανάκληση ενός διορισμού εισηγητή γίνεται διότι ο εισηγητής έχει παραβιάσει τους κανόνες συμπεριφοράς και το καθεστώς διαφάνειας και επομένως υπόκειται σε μια πολιτικού χαρακτήρα ή διοικητικού χαρακτήρα κύρωση, ενώ το ερετό αξίωμα είναι κάτι πιο βαρύ, πιο σημαντικό, το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με, την ίδια, με τον ίδιο τρόπο. Πρόεδρε, καλή σας μέρα. Νομίζω ότι με πολύ επιδεξιό τρόπο καταρτήσατε τους, ε, το θέμα της διαντολογίας, της συμπεριφοράς στο κανονισμό. Έχω όμως δύο-τρία σχόλια τα οποία θα ήθελα να σας παρουσιάσω. Θα το περιμένετε άλλωστε. Καταρχάς, για το θέμα του εισηγητή. Δεν νομίζω ότι είναι απαραίτητο να συμπληρώσουμε και να ενισχύσουμε τις κυρώσεις που έχουμε ήδη με επιπλέον κυρώσεις για να αποβάλουμε έναν εισηγητή από την Επιτροπή. Αν η Επιτροπή έχει την αίσθηση ότι ο εισηγητής έχει παραβιάσει τον κανονισμό, φυσικά θα απορρίψει και δεν θα δεχτεί την έκθεση. Νομίζω ότι μάλλον θα τα περιπλέξουμε τα πράγματα υπερβολικά. Αν ε, ορίσουμε επιπλέον κυρώσεις τέτοιου τύπου. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις ε, ομάδες της μικτές, στην τροπολογία 3, νομίζω ότι θα ήταν απαραίτητο οι λεπτομέρειες ε, οι οικονομικές σε ό,τι αφορά τις μικτές ομάδες να δημοσιεύονται δεν χρειάζεται να δημοσιεύονται στο διαδικτύο. Νομίζω ότι είναι επαρκές να ενημερώνονται οι κοσμήτορες. Και οι κοσμήτορες ε, με κάθε σεβασμό αν είναι εδώ στην αίθουσα. Κοιτάξτε, είναι λίγο σκοτεινό σώμα, να το πω έτσι, οι κοσμήτορες, άρα να δημοσιεύονται συγγνώμη, στο διαδίκτυο. Η διαφάνεια επιτάσσει να δημοσιεύονται αυτές οι πληροφορίες που λαμβάνουν οι κοσμήτορες στο διαδίκτυο. Για την τροπολογία 6, όπου αναφέρεται το θέμα της δεοντολογίας. Η αναφορά Το selflessness στα αγγλικά ακούγεται λίγο περίεργο. Ανιδιοτέλεια. Κάπως ευαγγελική θα έλεγα. Ως έννοια. Δεν νομίζω ότι αυτό ταιριάζει απόλυτα σε ένα τέτοιο κείμενο κανονισμού. Νομίζω όμω ότι το πρωτότυπο κείμενο ήταν στα γαλλικά γραμμένο. Δεν είδα τι λέει στα γαλλικά, αλλά ίσω θα μπορούσαμε να το δουλέψουμε με κάποιον ειδικό στην αγγλική γλώσσα για να βρούμε μια λιγότερο θρησκευτική, αν θέλετε, λέξη. Για να εκφράσουμε αυτό που θέλουμε. και αυτό που ζητάμε από τους βουλευτές. Τροπολογία 9. Να ρωτήσω το εξής. Πιστεύετε ότι θα μπορούσε να, υπήρ... να υπάρξει σύγκρουση ή τέλο πάντων προβλήματα μεταξύ της υποπαραγράφου Β, α, συγγνώμη, του 2Γ, όπου αναφέρεται ότι οποιαδήποτε αμοιβόμενη δραστηριότητα Ε, που συμπεριλαμβάνει και τους αυτοαπασχολούμενους θα πρέπει να δημοσιεύεται μεταξύ λοιπόν αυτής της παραγράφου Γ και μεταξύ της Ε που ορίζει ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα ορίζει ε, ένα όριο για τη συνολική αμοιβή που ανέρχεται στα 5.000 ευρώ ανα ημερολογιακό έτος. Ίσως να εξετάσουμε κατά πόσον υπάρχει απόλυτη σαφήνεια επ' αυτού. Μήπως υπάρχει κάποια αντίφαση μεταξύ των δύο παραγράφων, αλλά είναι σημαντικό να μην εισάγουμε κανόνες που θα προκαλέσουν περαιτέρω διαφωνίες. Και τέλος, για την τροπολογία 13 που αναφέρεται στην Επιτροπή Διοντολογίας ως συμβουλευτικό σώμα να διευκρινίσουμε νομίζω κατά πόσο η Επιτροπή αυτή Διοντολογίας μπορεί να προβεί σε ακρόαση του κατηγορούμενου αναφέρεται ότι ο πρόεδρος μπορεί να τον καλέσει. Αλλά δεν ορίζεται ποιες είναι οι αρμοδιότητες της Συμβουλευτικής Επιτροπής σε ό,τι αφορά τον εν λόγω, τον εν λόγω βουλευτή. Νομίζω προσωπικά ότι η Επιτροπή Διοντολογίας θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να καλέσει τον κατηγορούμενο σε ακρόαση. Αυτό θα πρέπει να ορίζεται όμως ρητά. Γιατί αν το αφήσουμε ανοιχτό, θα προκληθούν πολλά μελλοντικά προβλήματα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε και εισηγητά. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση η οποία λαμβάνει χώρα εδώ. Βλέπω ότι έχουν διαφορετικές απόψεις τα μέλη της Επιτροπής μας, τουλάχιστον σε, κάθε, σε κάποια λεπτομεριακά θέματα. προτού συνεχίσουμε λοιπόν τη συζήτηση. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι οι διαφορές αφορούν την τεχνική επίλυση των προβλημάτων. Αλλά γενικά επί της αρχής υπάρχει συμφωνία μεταξύ μας. Και εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι μια εξαιρετική. Η έκθεση του κ. Κασίνη είναι εξαιρετική. Επίσης είναι εξαιρετικό το έργο της ομάδας εργασία, Είναι τρίτη φορά που εγώ συμμετέχω σε μια τέτοια διαδικασία μετα, μεταρρύθμισης του κώδικα συμπεριφοράς των ε, ε, βουλευτών που έχουν σπηλωθεί ορισμένε φορές στο παρελθόν από πολιτικά σκάνδαλα οι υπολήψει του, και επομένως είναι απαραίτητο να μπορέσουμε να βρούμε σαφεί ε, εύστοχες αλλά και ισορροπημένες λύσεις για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά. Από την απόψη αυτή θέλω να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα κύριε Κασίνη. Εδώ δεν ε, εργαζόμαστε μονάχα για τους εαυτούς μας. Έχουμε ένα καθήκον να φέρουμε σε πέρας, το οποίο το ασκούμε με εντολή των εκλογέων μας και επομένως θα πρέπει να εξασφαλίσουμε και την εμπιστοσύνη τους. Αυτό είναι μια βασική αρχή της εργασίας μας και αυτό παραβιάζεται πολλές φορές όταν οι συνάδελφοι παραβιάζουν αυτή την αρχή και δεν δρούν ή δεν ψηφίζουν ακολουθώντας το συμφέρον των πολιτών, των εκλογέων τους, αλλά ακολουθώντας άλλα συμφέροντα, συμφέροντα τρίτων, όταν ακόμα προσπαθούν να αποκομίσουν και κάποια πλεονεκτήματα με το να έχουν μια συγκεκριμένη στάση σε μια ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ρόλο τους ως μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ιδιαίτερα ως εισηγητές, ως πρόεδροι επιτροπών κτλ. Αυτό σημαίνει κατάχρηση εξουσίας, κατάχρηση της υποχρέωσης να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα των πολιτών για τα οποία εξελέξαν κτλ. Αυτό φυσικά καταστρέφει την εμπιστοσύνη στους βουλευτές μας, μια εμπιστοσύνη η οποία μόνο με αργό τρόπο μπορεί να οικοδομηθεί και επομένως καταραίει εν μέρη και το οικοδόμημα του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας αν το επιτρέψουμε αυτό. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να κάνουμε κάτι για να εξασφαλίσουμε την επίτευξη μιας μεγαλύτερης διαφάνειας και τη ύπαρξη σαφών κυρώσεων. Γι' αυτό θα ήθελα να πω ότι έχουμε εξασφαλίσει βέβαια αυτήν την συνένεση μεταξύ μας για τις βασικές αρχές, αλλά όπως και ο Άντρου Λιγάκη έχω την εντύπωση ότι Χαίρομαι μεν ότι ο εισηγητής και πρόεδρός μας της Επιτροπής μας έχει κάνει μικρές προσθήκες και βελτιώσεις. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να δούμε ακριβώς ποιος είναι ο ρόλος ενός εισηγητή σε μια επιτροπή, γιατί όταν κάποιος αναλαμβάνει το έργο του εισηγητή, αυτό δεν το κάνει από τη δική του προσωπική έγκλη και εξουσία, είναι κάτι το, με το οποίο τον επιφορτίζει ένα κοινοβούλιο. Είτε είναι οι συντονιστές, είτε ένα πολιτικό κόμμα. Αυτή η ανάληψη λοιπόν του καθήκοντος του εισηγητή βασίζεται και στην εμπιστοσύνη της οποίας χαίρει από το σύνολο κοινοβούλιο. Επομένως θα πρέπει να συμπεριφέρεται με ένα τέτοιο τρόπο ο εισηγητής ώστε να μην καταχραστεί αυτή της εμπιστοσύνη. Αν λοιπόν κάποιος κάνει μια έκθεση σε ένα τομέα όπου είναι γνωστό και αποδείξιμο ότι έχει αποκομίσει κάποια πλεονεκτήματα από την δράση του από, από την πλευρά τρίτων, τότε αυτό πράγματι αποτελεί μια, ε, μια κατάχρηση. Τώρα, για το πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό των καταχρήσεων ε, και οι κυρώσει που πρέπει να επιβληθούν, εδώ δεν είμαι απόλυτα σίγουρος. Εσεί αναφέρεστε και σε άλλα αξιώματα μέσα στο Κοινοβούλιο, κύριο Κασίνη, αλλά όχι μονάχα αυτά που έχουν να κάνουν με την συγκεκριμένη Επιτροπή. Αναφέρεστε λοιπόν στο άρθρο 7 του τωρινού κώδικα συμπεριφορα όπου είναι η, Επιτροπή των, η Συνέλευση των Προέδρων, το 7 Δέλτα, που θα πρέπει να αποφασίσει υποβολή στην ε, ε, στην ε, συνέλευση των Προέδρων βάσει του 7 Δέλτα να ανακαλέσει το αξίωμα ενός εισηγητή από κάποιο βουλευτή. Εγώ αναρωτιέμαι όμως αν αυτό το, όργανο το οποίο είναι αυτό το οποίο δίνει την, διορίζει τον εισηγητή να είναι και αυτό το οποίο αφαιρεί το αξίωμα του εισηγητή. Εγώ συμφωνώ και με τον κύριο Σαλόμο, ο οποίος λέει ότι όταν πρόκειται για ένα ερετό αξίωμα το οποίο ανακαλείται, αυτό σημαίνει ότι είναι κάτι το οποίο αφαιρεί εξουσία και από τους πολίτες. Μια εκλεγμένη πολιτική θέση είναι ένα πρόσθετο καθήκον το οποίο δίδεται σε κάποιο άτομο και η ανάκληση αυτού του αξιώματος ε, συνοδεύεται και από μία ε, ουσιαστικά μείωση της, ε, της αξιοπρέπειας που έχει ένα άτομο ως πολίτης. Αλλά όταν δεν πρόκειται για αιρετά αξιώματα, όπως ε, αναφερθήκατε στην ε, περίπτωση της Ισπανίας, δεν μπορεί κανείς να αφαιρέσει βέβαια το αξίωμα του βουλευτή από κάποιο άτομο. Μόνο ένα δικαστήριο μπορεί να το κάνει ή μόνο οι εκλογείς στην επόμενη <clears throat> εκλογή. Αλλά μπορούμε σίγουρα να αφαιρέσουμε από ένα βουλευτή τις ε, ευθύνες και τα αξιώματα τα οποία έχει μέσα στο Κοινοβούλιο, όχι το ίδιο το αξιώμα του βουλευτή. Επομένως έχω μια διαφορετική αντιμετώπιση και επομένως συμπερασματικά. Καταρχήν συμφωνώ με την, ε, το περιεχόμενο της έκθεσης και θέλω να επενέσω και να ευχαριστήσω τον ε, εισηγητή γιατί έχει βελτιώσει σημαντικά το περιεχόμενο της ομάδας εργασίας. Πριν δώσω το λόγο στον συνάδελφο Σόντεργάρντε για να μπορέσω να προσανατολίσω τη συζήτηση γύρω από συγκεκριμένα στοιχεία. Το άρθρο 19 του κανονισμού λέει ότι, είναι, ότι πρόκειται για διαδικασία εφαρμογή των κυρώσεων. Η διάσκεψη των προέδρων μπορεί να αποφασίσει με τα τρία πέμπτα, ειδική πλειοψηφία δηλαδή, που εκπροσωπεί τουλάχιστον τρεις πολιτικές ομάδες, μπορεί λοιπόν να προτείνει στο Κοινοβούλιο την ανάκληση αξιωμάτων. Ποια αξιώματα, προέδρου, αντιπροέδρου, αντιπροέδρου επιτροπής, ε, ε, αντιπροσωπείας ή οποιοδήποτε άλλου αξιώματος ε, στο οποίο έχει εκλεγεί ο βουλευτής μέσα στο κοινοβούλιο. Η πρόταση πρέπει να εγκριθεί από το Κοινοβούλιο. Δεν αρκεί δηλαδή η διάσκεψη, του κοινο... η διάσκεψη των Προέδρων, αλλά χρειάζεται και η Ολομέλεια να εκφραστεί στα δύο τρίτα. Δεν μιλάμε λοιπόν εμείς για το για το εκλογικό αξίωμα όπως προκύπτει από τις εκλογές αλλά για την έμεση ανάθεση αξιώματος εντολής από την Ολομέλεια. Είναι σωστό αυτό το οποίο λέει εδώ ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί δηλαδή η ίδια ακριβώς διαδικασία και για την ανάκληση του ορισμού εισηγητή. Και θα πρέπει να πούμε ότι η διάσκεψη των προέδρων θα πρέπει να καλέσει την αρμόδια επιτροπή να ανακαλέσει τον εισηγητή, τον ορισμό του εισηγητού. Συγγνώμη. Ο κύριος Σόντεργάρντεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνώ με εκείνους που ανέφεραν ότι το θέμα στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι οι πολίτες να έχουν εμπιστοσύνη σε αυτούς που βρίσκονται εδώ στο Κοινοβούλιο. Δεν θα πρέπει να επιτρέπονται καταχρήσεις στις θέσεις αυτές για να δημιουργούνται οικονομικά συμφέροντα, να εξυπηρετούνται οικονομικά συμφέροντα. Και νομίζω ότι αυτό αποτελεί ένα από τα τεράστια προβλήματα εδώ στη συζήτηση, γιατί οι κυρώσεις που υπάρχουν σήμερα, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι υπήρξε παραβίαση του κώδικα διοντολογίας, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 153 δεν προκαλούν αρκετό φόβο αν θέλετε, δεν δρούν αρκετά ανασταλτικά. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά α, τις επαφές με τα λόμπι. Αν υπάρχει μια κύρωση 200 ευρώ, ε, εντάξει, δεν είναι και τόσο τρομερό το ποσό. Αντίθετα, για παράδειγμα με την ενδεχόμενη ε, ακύρωση αμοιβών για συγκεκριμένες ημέρες. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά το άρθρο 153. Το θέμα είναι η πολιτική κύρωση. Αυτό θεωρώ ότι ήταν πιο σημαντικό. Συζητήσαμε διάφορα ζητήματα με τον εισηγητή, αλλά τίφεται και το θέμα της δημοσίευσης. Το άρθρο 8 παράγραφος 5 τίθεται αυτό το θέμα. Θα πρέπει να δημοσιεύονται αυτά στην ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου. Νομίζω ότι είναι σημαντικό και θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι όλα αυτά θα, γίνονται θα πρέπει να γίνονται με απόλυτη διαφάνεια και στο, στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου. Δεν είναι δυνατόν. Μάλλον θα πρέπει να είναι να αρκετά να προβάλλονται αυτές οι πληροφορίες. Να είναι εύκολο να το βρει κανεί. Άλλο ένα πρόβλημα έχω όμως σε ό,τι αφορά το άρθρο 1 και 2. Δεν καταλαβαίνω την λογική δομή, αν θέλετε, των άρθρων. Όλα αυτά προέρχονται, ξέρετε, από την ομάδα εργασίας και αναφέρονται στο άρθρο 1 οι γενικές αρχές, στο δε άρθρο 2 ορίζονται οι βασικές υποχρεώσεις των βουλευτών. Κοιτώντας όμως την οπτική γωνία και για τα δύο αρχεία, και για τα δύο άρθρα, συγγνώμη, είναι η ίδια ουσιαστικά, γιατί αναφέρεται ότι στην άσκηση των καθηκόντων τους στα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι υποχρεωμένα και το καθεξής. Και στο άρθρο 1 και στο άρθρο 2 και παραθέτω κατά την εντολή και την άσκηση της εντολής του στα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υποχρεούνται να. Ε, άρα ποια είναι η διαφορά μεταξύ των γενικών αρχών όπως ε, ονομάζονται και των σημαντικών υποχρεώσεων καθηκόντων των βουλευτών. Στο άρθρο 2, έμα ε, και στις δύο περιπτώσεις για μια υποχρέωση μιλάμε. Εντάξει, μπορούμε να κάτσουμε να συζητάμε, αν θέλετε, τις υποχρεώσεις που αναφέρονται κατά πόσο είναι σκόπιμες ή όχι. Αλλά αυτό, κοιτάξτε, προέρχεται και από τις διάφορες παραδόσεις που υπάρχουν στις διάφορες χώρες. Εγώ, για παράδειγμα, δεν θέλω να, να υποχρεούμε να είμαι αμερόληπτος. Κοιτάξτε, εγώ προέρχομαι από ένα κόμμα. Από αυτό το κόμμα με εκλέξανε. Άρα δεν είμαι αμερόληπτος. Δεν έχω εκλεγεί ως πολιτικός για να είμαι αμερόληπτος. Δεν ξέρω αν με εξέλεξαν εδώ στο κοινοβούλιο για να εκπροσωπήσω το γενικό συμφέρον. Αλλά κοιτάξτε, είναι βέβαιος ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές στο πώς ε, οι συνάδελφοι ερμηνεύουν τον γενικό όρο γενικό συμφέρον. Είτε είναι κανείς από την αριστερά, από τη δεξιά, από, την, από το κέντρο του πολιτικού φάσματος. Νομίζω ότι θα έπρεπε να επικεντρωθούμε στα πιο ουσιώδη ζητήματα. Στα ζητήματα του πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε εμπόδια, να ορίσουμε κυρώσεις που θα αποτρέψουν το ενδεχόμενο κάποιος να δεχτεί χρήματα ή άλλα πλέον για να προασπίσει μια θέση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και κάτι τελευταίο που ήθελα να αναφέρω, το ποιος μπορεί να εκπληρώσει μία εντολή να καλέσει μία εντολή που έχει λάβει. Νομίζω. Σίγουρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί να ανακαλέσει μία εντολή η οποία έχει αποδοθεί από τους ε, εκλογείς. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε αποφασίσει και εμείς ήδη. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι έχουν επιλέξει κάποιον για να αναλάβει παραγωγή χάρη μια εισηγεσία είναι και αυτοί τα ίδια άτομα τα οποία θα πρέπει να ανακαλέσουν αυτή την εντολή. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στο να μην προκύψουν κίνδυνοι οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν μετά για να επιβληθούν ουσιαστικά πολιτικές κυρώσεις, να χρησιμοποιηθούν για πολιτική εκμετάλλευση. <clears throat> Πρέπει να υπάρξει μια συμφωνία στη συνέλευση των Προέδρων ή μέσα στην αρμόδια επιτροπή και να υπάρξει διαπίστωση ότι πράγματι κάποιος έχει πάρει ε, ωφέλη οικονομικά ή άλλα για να υποστηρίξει μια συγκεκριμένη πολιτική γραμμή. Αυτοί όμως οι οποίοι θα πρέπει να την πάρουν αυτή την ε, απόφαση για να ανακαλέσουν την εντολή είναι αυτοί που του έχουν δώσει την εντολή καταρχήν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Είναι εξαιρετική η έκθεση που έχουμε εδώ μπροστά μας. Νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό υπάρχει μεγάλη συμφωνία και είμαστε σε καλό δρόμο για την περιγραφή του κώδικα συμπεριφοράς. Ε, έχουμε το Μητρό Διαφάνειας και νομίζω ότι πέρσι κάναμε ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός προκειμένου να διαμορφώσουμε με πιο διαφανή τρόπο το Κοινοβούλιο κατέστη σαφής, ε, αναγκαίος μάλλον, ο κώδικας διοντολογίας, γιατί οι προηγούμενες ενέργειες ήταν πραγματικά εγκληματικής φύσεως. Απασχολούν τα δικαστήρια πλέον. Νομίζω ότι όλοι μας έχουν, έχουμε έναν δικό μας ε, πύχη διοντολογίας και το κοινό έχει το δικό του πύχη για τη συμπεριφορά των βουλευτών. Και αυτό μπορούμε λοιπόν να το καταγράψουμε, αλλά αυτό ποτέ δεν θα μας ε, προστατεύσει από μια ενδεχόμενη νέα τέτοια παραβίαση που θα φτάσει στα δικαστήρια από τα κοινοβούλια. Αυτό πρέπει να αποτρέψουμε και θα ήθελα να σας πω ότι εγώ δεν θέλω να κάνουμε ότι υπάρχει μια γενική υποψία. Να λέμε ότι αυτό στο παρελθόν πάντα ήταν δυνατόν και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και στην Επιτροπή Βιομηχανίας. Ξέρω πώς ε, διεξάγεται η νομοθετική διαδικασία και ξέρω τι όγκος δουλειάς υπάρχει. Και εγώ από την ομάδα μου πρέπει να σας πω ότι η δουλειά αυτή είναι πάρα πολύ περίπλοκη και είναι πάρα πολύ δύσκολο να εξευρεθεί συμφωνία και ομοφωνία σε νομοθετικές διαδικασίες. Θα πρέπει λοιπόν να προσέξουμε να μην δυσκολέψει υπερβολικά το έργο μας μόνο και μόνο επειδή στο παρελθόν κάποιοι δεν τήρησαν τους κανόνες. Αλλά αν ξεκινάνε εξωτερικά του Κοινοβουλίου τέτοιε διαδικασίε ε, προσαγωγή των ατόμων αυτών. Αυτό δεν είναι δουλειά του Κοινοβουλίου. Άρα, καλή είναι η διαφάνεια, αλλά θεωρώ ότι αυτό που είπε ο κ. Σομοντρικά ήταν πάρα πολύ θετικό να προσέξουμε να μην υπάρχει και πολιτική εκμετάλλευση σε ό,τι αφορά τις ε, κυρώσεις. Να προσέξουμε όταν ξεκινάμε και θέτουμε μια διαδικασία σε εξέλιξη, να προσέξουμε ποιο θα είναι το τέρμα της διαδικασίας αυτή, το τέλος της διαδικασίας. Αν ένας εισηγητής ε, ακολουθεί μια διαδικασία που δεν ε, ανταποκρίνεται στην άποψη της πλειοψηφίας, να μην υπάρχει δυνατότητα να εμποδιστεί. Άρα λοιπόν, Πρόεδρε, στα επτά σημεία νομίζω ότι ορίσατε και συνοψίσατε με πολύ καλό τρόπο πώς εμείς ως Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων μπορούμε να φανταστούμε το μέλλον της εργασίας αυτής και νομίζω ότι όσα προσθέθηκαν από την ομάδα εργασίας ήταν θετικά σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια και θα ήθελα εμείς ως ε, βουλευτές, ως αιρετοί εκπρόσωποι του κοινού να είμαστε και ορατή όντω στο κοινό και πρέπει να σας πω ότι 9% των 99% ε, των βουλευτών τηρούν αυτούς τους κανόνες, 99,9%. Και υπάρχει και ένα σύστημα πολιτικής υγιεινής εδώ στο Κοινοβούλιο, που λειτουργεί πολύ καλά. Είναι πολύ καλά λοιπόν αυτά που έχουμε γράψει, να τα εφαρμόσουμε, αλλά σας παρακαλώ να μην τα επεκτείνουμε, γιατί νομίζω ότι αυτό θα δυσκολέψει το έργο των ε, συναδέλφων που νομοθετούν. Αυτά περί Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι πολύ καλή ιδέα. Και υπάρχουν δυνατότητες ερμηνείας, όντως, αλλά είναι πολύ καλή η πρότασή σας, η οποία θα πρέπει να εφαρμοστεί το συντομότερο δυνατόν. Υπάρχει και ένα σχέδιο εφαρμογής και ελπίζουμε λοιπόν να ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή και μέσα από την Ολομέλεια μέχρι τα τέλη του έτους. Χωρίς μικρόφωνο πρόεδρος. Όχι, όχι, εσείς το ε, διακόψατε. Και με απόλυτο και με απόλυτο δίκαιο. <laughs> όλα, τα οποία γίνονται πια είναι, στο, είναι πολύ ε, ανοιχτά στην, ε, στα μέσα ενημέρωσης κτλ. Νομίζω ότι αυτό το οποίο πρέπει να κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι να τονίσει την δέσμευσή μας με τον κώδικα αυτό συμπεριφορά. Και θέλω να ευχαριστήσω και την ομάδα εργασία του Προεδρείου και εσά, κύριε Κασίλη για τον τρόπο με τον οποίο έχετε κάνει αυτή την ερμηνεία αυτών των ε, διατάξεων στον κανονισμό. Καταρχήν υπήρξε μια πολιτική προσέγγιση και είναι θετική και εμείς ως ομάδα του ΕΛΚ συμφωνούμε απόλυτα και την υποστηρίζουμε. Δεύτερον, και οι παρεμβάσει των συναδέλφων ήταν πολύ ενδιαφέρουσε και πλήρη περιεχομένου, γιατί αυτό είναι και ο σκοπό τη Επιτροπή μα να συζητήσουμε τα θέματα αυτά σε βάθο. Οι αμφιβολίε τώρα που προκάλεσαν τα πρώτα αυτά άρθρα στον κύριο Σέντεργατ εμένα δεν μου προξενούν πρόβλημα. Ποιον εκπροσωπούμε, αν εκπροσωπούμε συμφέροντα ή όχι. Οι Βρετανοί όταν ήταν καλοί Ευρωπαίοι σκεφτόντουσαν για όλα αυτά τα θέματα της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας με τον Blackstone και τον Burke θεωρώντας ότι δεν εκπροσωπούν μόνο τους εαυτούς τους αλλά, και το εκλογικό, αλλά καταρχήν το εκλογικό σώμα ο καθένας μπορεί να πιστεύει ότι θέλει σε κάθε πολιτικό κόμμα να εκπροσωπεί αυτό το οποίο νομίζει, αλλά όλοι μας σε τελική ανάλυση εκπροσωπούμε όλους, τα πάντα. Σε σχέση με τα ζητήματα τα οποία γέρθησαν εδώ πέρα. Θέλω καταρχήν να αναφερθώ στις αμφιβολίες που αναφέρατε εσείς ο ίδιος κύριε Πρόεδρε. Για τις διαπαραταξιακές ομάδες, τα intergroups. Εγώ ως πρόεδρος μιας διαπαραταξιακής ομάδας έπρεπε πάντα στην, ε, στη δήλωση συμφερόντων μου να καταγράφω αν αυτή η διαπαραταξιακή ομάδα μου έδινε κάποια υποστήριξη, γραμματιακή κτλ. Όλα αυτά είναι, στο, είναι σε δημόσια γνώμη, σε, είναι γνωστά, πάση Βρίσκονται στο ίντερνετ του Κοινοβουλίου. Εγώ πιστεύω ότι είναι σημαντικό το έργο των διαπαραταξιακών ομάδων Υπάρχουν πολλοί στο Κοινοβούλιο που κάνουν ό,τι μπορούν για να τροχοπεδίσουν το έργο των διαπαραταξιακών ομάδων. Αλλά η δημιουργία αυτών των ομάδων ήταν ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο για να μπορέσουμε να επιζητήσουμε τη συνένεση σε πολλά θέματα. Αν έχουμε λοιπόν την ευκαιρία να ακούσουμε τις απόψεις των μεν και των δε και να συζητήσουμε, αυτό είναι πολύ θετικό. Γι' αυτό η μεγαλύτερη διαφάνεια σημαίνει να υποστηρίξουμε και αυτές τις διαπαραταξιακές ομάδες, τα intergroups. Επίσης, ε, κύριε Πρόεδρε, Αναφερθήκατε στο θέμα της κύρωσης για κάποιο βουλευτή ο οποίος είναι εισηγητής αλλά δεν σέβεται τον κώδικα συμπεριφοράς. Εδώ υπάρχει και μία πτυχή που είναι σημαντική, που είναι το παιδαγωγικό στοιχείο, είναι το παράδειγμα το οποίο θέλουμε να δείξουμε. Αν θέλουμε να τονίσουμε ότι ένας βουλευτής δεν αξίζει να είναι πλέον εισηγητής, Νομίζω ότι αυτό πρέπει να το κάνουμε με τρόπο ο οποίος θα είναι πρόδειλος, θα είναι σαφής. Ο Άντριου Ντάφ ξεκινά από μια πιο πραγματιστική στάση που λέει εντάξει, του καταψηφίζουμε την έκθεσή του και επιτυχάνουμε τελικά το στόχο. Αλλά στην πραγματικότητα η πρακτική σημαίνει ότι οι συγητές είναι προϊόν, η ενός είναι προϊόν συμφωνίας των συντονιστών βάσει του καβαλιστικού συστήματος των μορίων. Αλλά στη συνέχεια η πρόταση αυτή υποβάλλεται στην αρμόδια επιτροπή. Λένε ότι ο ΤΑΔΕ προτείνεται ως εισηγητής. Είναι η ίδια η κοινοβουλευτική επιτροπή η οποία τον εγκρίνει. Μπορεί να θεωρήσει όμως ότι αυτό το άτομο δεν είναι το κατάλληλο. Υπάρχει η μία έγκριση λοιπόν από την κοινοβουλευτική επιτροπή γι' αυτό. Πιστεύω ότι το λογικό σε αυτήν την περίπτωση θα ήταν ότι αυτός ο οποίος έχει επιλέξει κάποιον ως εισηγητή να είναι αυτός ο οποίος μπορεί να αποσύρει την εμπιστοσύνη του σε περίπτωση που υπάρχει μια παραβίαση του κώδικα συμπεριφορά. Γι' αυτό θα ήμουν υπέρ του να είναι η αρμόδια επιτροπή η οποία ενδεχομένως μετά από κάποια ένδειξη ενδεχομένω της συνέλευσης των Προέδρων κάνει την ε, απόσυρση της εντολής του εισηγητή. Κάτι άλλο τώρα, δεν ξέρω αν σύμφωνα εδώ με τον κύριο Νταφ. Νομίζω ότι αυτή η Συμβουλευτική Επιτροπή είναι σημαντική, όπως είπε και ο κύριος Γκερέρο, γιατί υπάρχουν πολλές περιπτώσεις προσωπικού χαρακτήρα που μπορεί να μην είναι τόσο σαφής. Ξέρω την ε, δική μου, από τη δική μου εθνική εμπειρία στο Ισπανικό Κοινοβούλιο ότι υπήρξαν πολλές περιπτώσεις όπου δεν ξέρει κανείς αν το να είναι ένας βουλευτής ε, μέλος κάποιου διοικητικού συμβουλίου μιας εταιρείας αποτελεί ασύμβατο ή ασυμβίβαστο με το αξίωμα του βουλευτή ή δημιουργεί προβλήματα. Εγώ πιστεύω ότι οι κανόνες που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ιδιαίτερα προεδρικού χαρακτήρα. Τα αφήνει όλα στα χέρια του Προεδρού του Κοινοβουλίου. Εγώ νομίζω ότι ο βουλευτή, όταν υπάρχει μια ευλογή αμφιβολία σε σχέση με το αν εμπίπτει η περίπτωσή του σε αυτά τα οποία λέει ο κανονισμό, θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να ακουστεί η άποψή του από τη Συμβουλευτική Επιτροπή και όχι μονάχα από τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου. Ο Πρόεδρο ούτω ή άλλω είναι πολύ άσχολος, έχει κάποια πολιτικά καθήκοντα. Νομίζω ότι αυτή η Συμβουλευτική Επιτροπή είναι πιο αρμόδια για να ακούσει την άποψη ενός βουλευτή και να δώσει μια γνωμοδότηση στη συνέχεια στον πρόεδρο του Κοινοβουλίου. Συνολικά λοιπόν με όλα αυτά θα ήθελα καταρχήν φυσικά να σας ευχαριστήσω για το έργο σας και να τονίσω ότι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα είναι στη διάθεσή σας για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε περαιτέρω αυτό το κείμενο το οποίο νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή θετική είδηση σε στιγμές που όπως είπε και ο κύριος Γκερέρο οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν αρκεί να είμαστε έντιμοι όπως η γυναίκα του Κέσσα αλλά πρέπει να φαινόμαστε και έντιμοι. Και όσο πιο πολύ δείχνουμε ότι είμαστε έντιμοι, τόσο καλύτερο. Τόσο καλύτερο. Ευχαριστώ κύριε Μέντες, ο κύριος Μπρόνς. Μπορεί να μην είμαι ο πρώτος που θα υπερασπιστώ τη θύμη του Κοινοβουλίου, αλλά είναι φυσικά σημαντικό όλα τα δημόσια αξιώματα να ε, διεξάγονται με τιμιότητα. Και αυτό ισχύει και για το Κοινοβουλίο μας και για άλλα κοινοβούλια. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να κάνουμε διάκριση μεταξύ των ε, βουλευτών που συνειδητά παραβιάζουν τους κανόνες και είναι διεφθαρμένα και όσους ε, ε, λόγω ε, σύγχυσης, αν θέλετε, ή οριακών καταστάσεων παραβιάζουν κάποιες υποχρεώσεις. Στην τροποποίηση 9, στην οποία αναφέρθηκε και ο κ. Νταφ προηγουμένως, στο 9 ε αναφέρεται ένα ποσό. Αν υπερβαίνεται το ποσό των 50, το 5.000 ως αμοιβή. Αλλά στο γάμα, στο 9 γάμα γίνεται αναφορά σε οποιαδήποτε αμοιβόμενη δραστηριότητα, ακόμα και σε μικρή αμοιβόμενη δραστηριότητα. Στο 9H αναφέρεται οποιοδήποτε, στο Z αναφέρεται οποιαδήποτε οικονομική υποστήριξη. Και οποιαδήποτε οικονομικά συμφέροντα στο ΙΤΑ. Όλοι φυσικά μπορούμε να πούμε ότι δεν επηρεαζόμαστε από οικονομικά συμφέροντα, αλλά θεωρώ ότι η σύγχυση θα μπορούσε να διαλυθεί ορίζοντας ρητά το τι συμπεριλαμβάνεται και τι δεν συμπεριλαμβάνεται. Και επίσης με πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις στις οποίες θα πρέπει να απαντάν οι εν λόγω βουλευτές προκειμένου να μην υπάρχει δικαιολογία ότι δεν κατάλαβε σε περίπτωση που υπάρχει συγκεκριμένη ερώτηση. Είναι ωστόσο επικίνδυνο να θέσουμε και να κατηγορήσουμε αν θέλετε κάποιους ε, αθώους οι οποίοι θα μπουν και θα πέσουν σε μια πολιτική παγίδα ενδεχομένω. για να το θέσω ε, έτσι. Ευχαριστώ. Ζήτησε και πάλι το λόγο για να ολοκληρώσει ο κύριος Γκερέρο. Πάρα πολύ σύντομα για να μην υπάρχει σύγχυση για τη θέση της σοσιαλιστικής ομάδας. Εγώ συμφωνώ με τον κύριο Χέφνερ και με τον πρόεδρο σχετικά με το θέμα των εκλεγμένων αξιωμάτων υπήρξε ένα λάθος από τη μεριά μου, είχα κάνει λάθος τον όρο. Ευχαριστώ κύριο Σέπλινγκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να σα ευχαριστήσω και για αυτή την έκθεση. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση. Έχω ορισμένε σκέψει να σα υποβάλω. Η πρώτη αφορά την συμβουλευτική αυτή επιτροπή. Η τροπολογία 12 είναι αυτή στην οποία αναφέρομαι. Ένα ερώτημα μονάχα είναι αυτός ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπίσουμε ζητήματα ε, διαφάνειας όταν κάποιος ε, θα πρέπει να διορίζεται και όχι να εκλέγεται. Όταν κάποιος διορίζεται και όχι εκλέγεται. Είναι ο τρόπος με τον οποίο θα αυξήσουμε την νομιμοποίησή μας στα μάτια του πολίτη. Μήπως θα πρέπει αυτό το σώμα να εκλέγετε και όχι να διορίζετε γιατί αλλιώς φαίνεται ότι κάπου έχει ειδικά προνόμια. Δεύτερον, και μετά έρχομαι στο ερώτημα ποιος, φυλά, ποιος μας φυλάσει από τους φύλακες. Ποια θα είναι η διαδικασία αυτής της ε, Συμβουλευτικής Επιτροπής. Θα είναι δημόσια τα απεπραγμένα τους, οι αποφάσεις τους, οι σκέψεις τους, θα καταγράφονται κάπου. Θα δημιουργούν κάποιο προηγούμενο. Αυτό ίσως δεν είναι λάθασμένη λύση, γιατί εδώ έχουμε προβλήματα αμφισημίας τα οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Είναι προβλήματα τα οποία θα επανέλθουν εξάλλου. Και είναι δεσμευτικέ οι αποφάσει αυτή τη Συμβουλευτική Επιτροπή. Θα πρέπει να ξέρουμε αν υπάρχει δεσμευτικό χαρακτήρα ή όχι σε αυτά που αποφασίζει η Επιτροπή αυτή. Και επιπλέον στην τροπολογία 8. Χωρί μικρόφωνο ο κύριο Μέντες Δεβίγο. Η τροπολογία 8 σε περιπτώσεις αμφισημίας μπορεί το εμπλεκόμενο μέλος να ζητήσει τη γνωμοδότηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής. Εκεί πρέπει να υπάρχει και μια υποχρέωση Συμβουλευτικής Επιτροπής μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα 30 μέρες, 15 μέρες να απαντήσει. Όχι να το αφήσουμε στον αέρα ότι α, κάποτε θα δώσουν μια απάντηση. Πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι στο θέμα αυτό. Και το άλλο θέμα αφορά τα οικονομικά συμφέροντα και τα συναφή. Εδώ νομίζω θα πρέπει να είμαστε πιο σαφείς, να καθορίσουμε με ευρύτερο τρόπο τα οικονομικά συμφέροντα και αναφέρομαι στην τροπολογία 9 τώρα. Ο δημόσιος τομέας και ο ιδιωτικός τομέας που μια φορά και ένα καιρό ήταν σαφώς ξεχωριστή. τώρα πια δεν είναι. Υπάρχει μεγάλη επικάλυψη μεταξύ των δύο περνάνε από το δημόσιο στο ιδιωτικό τομέα με μεγάλη ευκολία τα άτομα όπως αλλάζουν πουκάμισο και χρησιμοποιούν την εμπειρία που έχουν αποκομίσει στον ένα τομέα για να τις χρησιμοποιήσουν στον άλλο. Μήπως πρέπει να βρούμε τρόπο, κάποιο τρόπο να περιλάβουμε και την υπηρεσία σε κάποια κυβερνητική υπηρεσία. Γιατί και αυτή μπορεί να οδηγήσει στο να προσποριστεί κάποιος κάποιο πλεονέκτημα τοπικές ε, αρχές αυτοδιοίκησης, ε, κρατικές υπηρεσίες ή μη κυβερνητικές ΜΚΟ, κυβερνητικές ΜΚΟ κτλ. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Δεν πρόκειται μόνο για τον ιδιωτικό τομέα, είναι και ο δημόσιος τομέας ο οποίος και αυτός μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα, γιατί είναι το θέμα της εξουσίας, της εμπιστοσύνη, της διαφάνειας. Και πολλές φορές αυτά που έχει κάνει κανείς όταν έχει δουλέψει σε κάποιο δημόσιο τομέα είναι εξίσου σημαντικά με αυτά που έχει κάνει στον ιδιωτικό τομέα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βίλαντ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς ε, να αναφερθώ στη συνάδελφο Γκρότε και κατά στη συνάδελφο Μπόντς. Θα ήθελα λοιπόν να πω σαφώς ότι το έγγραφο αυτό το υποστηρίζω επί της αρχής και σίγουρα μπορούμε να συζητήσουμε για διάφορες γενικές αρχές και για άλλους όρους. Νομίζω ότι μετά από λίγο χρόνο θα προκύψουν και κάποιες λύσεις. Αλλά να αναφερθώ συγκεκριμένες τροπολογίες 19 και 12. Να πω ότι στα 14 χρόνια ποτέ δεν γνώρισα ούτε μία περίπτωση όπου κάποιος γλωμπιίστας με προσέγγισε και είπα ότι υπήρχε ακόμα και από μακριά δυνατότητα να υπερβώ τα όρια, να ξεπεράσω τα όρια. Άρα νομίζω ότι στις περιπτώσεις που μας απασχολούν εδώ, οι συνάδελφοι οι οποίοι έκαναν τις παραβιάσεις ήταν επιλεγμένοι. Άρα νομίζω ότι δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και κάποια άλλα ε, ζητήματα σε ό,τι αφορά το έγγραφο αυτό. Αν υπάρχουν λοιπόν κάποιοι προκλητικοί παράγοντες εδώ στο Κοινοβούλιο, θα πρέπει να τιμωρούνται. Καταρχάς, αλλά θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και αυτούς που βρίσκονται από την άλλη πλευρά του Κοινοβουλίου. Δηλαδή, αν είχα λάβει εγώ κάποια τέτοια πρόταση, θα είχα πει πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η πρότασή σας, αλλά θα είχα πάει στη συνέχεια και στον πρόεδρο να το καταγγείλω. Και άρα έτσι θα πιάναμε και αυτούς που παραβιάζουν τους κανόνες μας από έξω. Το 95% είπε ο κύριος Σόνδεργκάρτε ε, εργάζονται τίμια ή αυτό προσπαθούν τουλάχιστον. Και νομίζω ότι αυτές τις περιπτώσεις δεν θα πρέπει να τις δημοσιεύουμε στην ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου. Νομίζω ότι τα καλά θα πρέπει να δημοσιεύουμε, αν και τα κακά μαντάτα γίνονται γνωστά από μόνα τους και οι σχετικοί σύνδεσμοι. Να αναφερθώ τώρα στον Πρόεδρο. Νομίζω ότι σε ό,τι αφορά το άρθρο 19 και 12 δεν έχουμε ολοκληρώσει την εργασία μας. Θα χρειαστεί και μια κουλτούρα, αν θέλετε, της εφαρμογής της ε, συμβουλευτικής αυτής επιτροπής, που είναι κάτι καινούριο. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να δραστηριοποιείται μόνο σε περίπτωση υποτιθέμενης ε, παραβίασης. Δεν θα πρέπει να δίνει μόνο βοήθεια κατευθυντική, αν θέλετε, το οποίο είναι δύσκολο, δύσκολα κατανάητο. Αν έρχεται ένα μέλος του Κοινοβουλίου και μας λέει ότι κοιτάξτε, έχω αυτή την κατάσταση, πώς να συμπεριφερθώ. Να πούμε ότι κοιτάξτε, πιστεύουμε ότι μάλλον προς αυτή την κατεύθυνση ψηφίσαμε και αποφασίσαμε γιατί ο βουλευτής αυτός θα βρεθεί θύμα της δημόσιας κοινή γνώμης αν τελικά δεν αποτεχθεί σωστή αυτή η σύσταση. Όχι, οι βουλευτές χρειάζονται σαφήνεια, χρειάζονται νομική βεβαιότητα. Άρα θεωρώ ότι θα έπρεπε να είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής αυτής, της Συμβουλευτικής Επιτροπής αυτής, να κρίνουν με απόρριτο χαρακτήρα και τη συμπεριφορά τρίτων εκτός κοινοβουλίου. Κάτι άλλο που με λυπεί ιδιαίτερα. Στο άρθρο 4, τροπολογία 9. Υπάρχει, ε, υπάρχουν πάρα πολλές ε, αόριστες νομικές ε, έννοιες. Τι είναι δηλαδή το όργανο διευθύνσης διαχείρισης. Δηλαδή η Συμβουλευτική Επιτροπή αναγνωρίζει ε, την Επιτροπή και το όργανο στο οποίο συμμετέχει κάθε βουλευτή ω διευθυντικό όργανο. Πρόκειται για μια αόριστη νομική έννοια. Και δεν δημιουργεί αυτονομική σαφήνεια και για την ε, Συμβουλευτική Επιτροπή. Και αυτό αποβαίνει ει βάρο και της επιτροπή, αλλά και του βουλευτή που αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα, μια βέβαιη κατάσταση. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα εισοδήματα, τα τακτικά ή μη, θεωρώ ότι η διατύπωση δεν είναι αρκετά σαφής και υπάρχει μεγάλο περιθώριο σύγχυσης. Για την τροπολογία 10 θα ήθελα να κάνω επίσης ένα σχόλιο. Η προφανής αξία, και αυτό με εκνευρίζει ιδιαίτερα. Δηλαδή τώρα τι είναι προφανές. Αυτό επιβαρύνει τον βουλευτή. Αυτός καλύτερα να το κρίνει. Δεν θεωρούμε ότι είναι προφανές, αλλά ποιος ξέρει. Θα ήθελα μία τιμή αγοράς. Κάτι τέτοιο να αναφέρεται κάποια φορά μου είχαν δώσει ένα πίνακα. Τι να σας πω, αυτή η αγορά, α, η τιμή αγοράς του πίνακα αυτού, της εικόνας αυτής, τι να σας πω, μπορεί να είναι μηδενική γιατί κανείς δεν θέλει να το αγοράσει, αλλά μπορεί να είναι και 2.000 ευρώ αν χρειαστεί. Τι να σας πω, θα ήθελα μεγαλύτερη σαφήνεια, θα ήθελα να προσταθεί μια παράγραφος 3. Γιατί αν ε, οριστεί ότι υπάρχουν δώρα τα οποία δεν μπορεί να αρνηθεί κανείς, αλλά έχουν μια αντικειμενική αξία. Το Γερμανικό Κοινοβούλιο ορίζει ότι ορίζει ότι αν δίδεται κάποιο δώρο, ορίζεται ως όριο τα 150 ευρώ και στη άλλη περίπτωση δεν πρέπει να το επιστρέψει, σε, εκτός κι αν χορηγήσει και πληρώσει την επιπλέον αξία πέρα από τα 150 ευρώ. Φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρησιμοποιεί ο τύπος. Και σε περίπτωση που λάβει κανείς τέτοια δώρα, δεν μπορείτε να πετάξει καν υπό απόλυτο απόδειτο πρέπει να τα πετάξει κανείς αυτά τα δώρα. Τέλος, Πρόεδρε. Θα ήθελα στις και σκέψεις να απευθυνθεί μεγαλύτερη έκκληση στις ε, συνηθισμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται. Χρειαζόμαστε δικαίωμα ασυλίας. Αν κατηγορείται για κάτι ένας βουλευτής και αν όντως κατά το εθνικό δίκαιο είναι ποινικό, ποινικά διώξιμο αυτό που έπραξε, αλλά αν δεν είναι αξιόπινη η πράξη του στο εθνικό δίκαιο, δεν υπάρχουν ε, κανονισμοί για το κάθε πόσο μπορούμε για παράδειγμα να ερευνούμε τα γραφεία των βουλευτών και έχουμε δυσκολευτεί στο παρελθόν και με την Όλαφ, με θέματα ασυλίας. Ένας από τους βουλευτές ε, παρατήθηκε κατευθείαν και δεν μιλάω μόνο για περιπτώσεις ε, βουλευτών που είχαν πάρει χρήματα, μιλάω και για άλλες περιπτώσεις, γιατί υπάρχουν απόρριτα έγγραφα τα οποία προστατεύονται από το δικαίωμα της ασυλίας. Άρα χρειάζεται να γίνει ένα σημαντικό βήμα σε ό,τι αφορά την ασυλία και εδώ θα ήθελα να απευθυνθεί μια τέτοια έκκληση στα όργανα αυτά που συμμετέχουν σε ετολογικές σκέψεις σε ό,τι αφορά θέματα ασυλίας. Eh, Ευχαριστώ. Ο κύριος Μέσσερσμιτ. Ε, Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, πρώτα απ' όλα θέλω να εστιάσω την παρέμβασή μου στην αρχή της διαφάνειας. Μπορεί να υπάρχει μια προληπτική δράση από τη δική μας πλευρά προληπτική και όχι κατασταλτική εκ των υστέρων. Δεν έχει νόημα στη συνέχεια να βάζουμε τους βουλευτές να πληρώνουν πρόστιμο οτιδήποτε τέτοιο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα της διαφάνειας. Αν έχουμε λάβει λοιπόν μια απόφαση που λέει ότι έχουν παραβιαστεί κάποιες αρχές διοντολογίες... Νομίζω ότι είναι προ το γενικό συμφέρον αυτό να γίνει γνωστό το ταχύτερο δυνατό. Αν θέλουμε οι κανόνε αυτοί να επηρεάσουν πράγματι τη συμπεριφορά των κοινοβουλευτικών κατά τη διάρκεια τη άσκηση τη εντολή του, η δημοσιότητα είναι η πιο αποτελεσματική κύρωση, δηλαδή να γνωρίζουν οι εκλογείς των βουλευτών αυτών ότι παραβιάστηκε ο κανόνα δεοντολογίας των βουλευτών. Νομίζω ότι μια απόφαση δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να ληφθεί. Βέβαια, αυτό η γνωστοποίηση, δημοσίευση δεν σημαίνει ότι μπορούν να δημοσιευτούν κάθε είδους λανθασμένες πληροφορίες, αλλά είναι απαραίτητο να υπάρχει ταχεία δημοσίευση. Ένα από τα πλεονεκτήματα της δημοκρατίας είναι ακριβώς το να μπορεί ο, βουλε... ο πολίτης να έχει τις πληροφορίες για τον βουλευτή του. Όπως ελέγχθη λοιπόν θα ήταν πολύ θετικό να έχουμε <clears throat> και τον θετικό και τον αρνητικό ορισμό μέσα στον κώδικα συμπεριφοράς, όπως ζητούν οι τροπολογίες 6 και 7. Να υπάρχει λοιπόν και η θετική δήλωση του τι κάνει ένας, τι κάνει ένας βουλευτής και αρνητική του τι δεν μπορεί να κάνει. Έχω όμως το εξή πρόβλημα για την τροπολογία υπαριθμών 7 για το άρθρο 2β. Εκεί αναφέρεται το θέμα της διαφθοράς. Όπως είπε και ο προλαλής σας, η διαφθορά είναι κάτι το οποίο σύμφωνα και με τους εθνικούς κανόνες είναι κάτι το οποίο αντιβαίνει στην νομοθεσία. Είναι... Υπάρχουν ίσως 27 διαφορετικές αντιμετωπίσεις της διαφθορά στα κράτη-μέλη μας. Είναι οι κανόνες των εθνικών κοινοβουλίων και των εθνικών δικαστηρίων που τελικά θα είναι αποφασιστικές. Μπορούμε να έχουμε δύο άτομα τα οποία έχουν εκλεγεί σε δύο διαφορετικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάνουν το ίδιο ακριβώς αδίκημα. Ένα από αυτά τα άτομα βάσει των εθνικών κανόνων υφίσταται κυρώσεις και, και χάνει το περδίεμ του στη συνέχεια, ενώ ο άλλος χάνει την ασυλία του και τον πετάνε στη φυλακή για το ίδιο αδίκημα. Αυτό είναι πραγματικά πολύ παράξενο πρέπει να καθορίσουμε ακριβώς τι εννοούμε όταν μιλάμε για διαφθορά. Και να πούμε ότι αυτό θα πρέπει να σημαίνει και απώλεια του δικαιώματος ενός βουλευτή να κάνει ορισμένα πράγματα μέσα στο κοινοβούλιο. Η διαφθορά θα πρέπει να σημαίνει την άρση της ασυλίας και μετά μόνο τα δικαστήρια μπορούν να πάρουν μια απόφαση σε σχέση με τα άτομα αυτά. Εάν εμείς όμως προστατεύσουμε αυτούς τους βουλευτές με το να αφαιρέσουμε μονάχα την ημερήσια αποζημίωσή τους, αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Πρέπει λοιπόν όταν υπάρχει και μία οποιαδήποτε υποψία για διαφθορά να έρεται η ασυλία και να παραπέμπεται το θέμα αυτό των εθνικών δικαστήριων. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο για μένα είναι καταφανές είναι το εξής. Αν αυτή η Συμβουλευτική Επιτροπή η οποία θεσπίζεται αποφασίζει να αφαιρέσει ημερήσει αποζημιώσει από κάποιο βουλευτή, θα είναι στη συνέχεια οι συντονιστές που θα αποφασίσουν ότι κάποιος πάβει να είναι εισηγητή. και θα πρέπει να πάρει την ε, εισηγεσία κάποιο άλλο ή κάποια άλλη πολιτική ομάδα ή αυτό θα πρέπει να εναπόκειται στις ίδιες πολιτικές ομάδε Νομίζω ότι αν κάποιο ορίζεται εισηγητή από του συντονιστέ, αν δεν μπορεί να είναι πια, να είναι πια εισηγητής, θα πρέπει το θέμα αυτό να παραπευθεί και πάλι στους συντονιστές και όχι να αποφασίσουν οι πολιτικές ομάδες ποιος θα τον αντικαταστήσει. Και κλείνω με ένα θετικό μήνυμα ότι υπάρχουν πολλά στοιχεία μέσα στην έκθεση του Πρόεδρου μας που είναι θετικά και μπορούν να υποστηριχθούν από εμά. Όταν πρόκειται πάντως για το θέμα της άρσης, της ασυλίας, ή της, ή της ε, αφαίρεσης ε, ημερησίων αποζημιώσεων χρειάζεται μια μεγαλύτερη σαφήνεια στο κείμενο αυτό. Ο κύριος Χέφνερ. Ήθελα εν συντομία να επανέλθω στο βασικό αυτό το θέμα του πώς αντιμετωπίζουμε τους εισηγητές. Για να είμαι ειλικρινή, καθόμουν και το σκεφτόμουν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, αν σωστά καταλαβαίνω. Αρχικά στο άρθρο 7 της ομάδας εργασίας είχαμε δύο διαφορετικές διαδικασίες επιβολής κυρώσεων. Η πρώτη ήταν ε, τα σημεία α ως δ, όπου αποφασίζει ο πρόεδρος ουσιαστικά και καθοριστικά και στην περίπτωση ε μόνο, όπου πρόκειται για την αφαίρεση των δικαιωμάτων των πολιτικών, ε, εκεί με τρία πέμπτα πλειοψηφία αποφασίζει η διάσκεψη των Προέδρων και μετά η Ολομέλεια με δύο τρίτα υποστηρίζει ή όχι την κύρωση αυτή. Αυτά ισχύουν σήμερα. Το πρόβλημα είναι το εξή. Η ερώτηση που έθεσε ο Πρόεδρος Καζίνη είναι πού θα ενταχθούν όλα αυτά. Και το θέμα θα ήταν ουσιαστικά όπως και τα υπόλοιπα αξιώματα θα έπρεπε να τα αντιμετωπίσουμε. Ωστόσο, το... η αίσθησή μου είναι για το που μπορούμε ακριβώς να τα εντάξουμε αυτά, ότι φυσικά αυτό αποτελεί ένα πάρα πολύ ψηλό εμπόδιο το οποίο έχουμε ορίσει και παρόλα αυτά Εξετάζοντας αυτά τα δύο συστήματα, αυτές τις δύο διαδικασίες που ίσχυαν ως τώρα, θα το αντιμετωπίσουμε όπως προτείνει ο πρόεδρος Καζίνης σαν ένα οποιοδήποτε άλλο αξίωμα. Εγώ όμως θεωρώ ότι το να μπορεί να αποφασίζει ο πρόεδρος μόνος του δεν πρέπει να αφορά τέτοια ζητήματα όπως για παράδειγμα η αφαίρεση η καθαίρεση ενός βουλευτή δεν μπορεί να αποτελεί τέτοιο θέμα που να αποφασίζει ο πρόεδρος μόνος του. Νομίζω ότι από πλευράς ε, βαρύτητας είναι πιο σοβαρή αυτή η κύρωση. Τα υπόλοιπα θέματα και αυτό που έθιξε ο κύριος ε, <laughs> Βίλαντ. Ε, χαίρομαι που ανησυχείτε για το αυξανόμενο όγκο απορριμμάτων στο Κοινοβούλιο και για τα δώρα αυτά που καταλήγουν και φυσικά δεν θα πρέπει να καταλήγουν εκεί και πώς θα πρέπει να γίνονται όλα αυτά με νομίμως καθαρό τρόπο. Όλα αυτά που λέτε είναι σωστά. Αλλά ζήτησα το λόγο επίσης άλλη μια φορά γιατί μου κάνει εντύπωση ότι στη συζήτηση αυτή κάνουμε και μία συζήτηση για την ιδιότητά μας και για τα αυτονόητα ως βουλευτές. Να κάνω λοιπόν μία παρατήρηση προς τον συνάδελφο Ζόντεργκαρτ και ελπίζω να με συγχωρέσατε γιατί αυτό που είπατε στην πρώτη, στο πρώτο τμήμα της εισήγησής σας είπατε ότι δεν εκπροσωπείτε το γενικό συμφέρον, εκπροσωπώ ένα συγκεκριμένο κόμμα και συγκεκριμένα συμφέροντα. Αυτά με ενόχλησαν γιατί αυτή η ιδέα του Κοινοβουλίου είναι ότι όλοι έχουμε διαφορετικές οπτικές γωνίες αλλά ότι αυτό είναι υπέρ του γενικού συμφέροντος. Έχουμε φιλελεύθερους κομμουνιστές και έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα. Αλλά ελπίζω παρόλα αυτά ότι όλοι να μην κοιτάμε ποιο είναι το δικό μας συμφέρον, ποιο είναι το συμφέρον της εκάστοτε ομάδας, αλλά ποιο είναι το κοινό συμφέρον. Γιατί, εξ όσων έχω καταλάβει για τον κομμουνισμό, δεν ισχύουν αυτά που λέτε. Και αυτό λοιπόν ήθελα να υπογραμμίσω. Ο κύριος Τέιν. Η κυρία Πάρα πολύ σύντομα θα λάβω το λόγο. Γιατί εγώ μπορώ να συμφωνήσω με αυτά που είπε ο κύριος Βίλαντ σε ό,τι αφορά τη χρήση ορισμένων νομικών ενιών. Και θέλω επίσης να αναφερθώ και σε δύο σημεία. Και για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό η Συμβουλευτική Επιτροπή να δώσει μονάχα μια γενική κατεύθυνση όχι μόνο συγγνώμη, να δώσει μια γενική κατεύθυνση, αλλά να δημιουργήσει και μια νομική ασφάλεια για το εμπλεκόμενο μέλος. Και για την τροπολογία 12 σε ό,τι αφορά τα δώρα. Εγώ έρχομαι από μια μικρότερη πολιτική ομάδα. Πολλές φορές κάνω παρουσιάσεις και ομιλίες στη Γερμανία. Πολλές φορές θα πρέπει να μείνω σε ένα μέρο που δεν είναι η, η εκλογική μου περιφέρεια. Και ξέρετε, ότι αυτά τα, το κόστος διανυκτέρευσης πολλές φορές το επομίζεται ο διοργανωτής μιας ε, εκδήλωσης. Όταν είσαι σε ένα ξενοδοχείο πεντάστερο στη Γερμανία, σίγουρα αυτό ξεπερνάει το όριο των 150 ευρώ πολλές φορές. Μπορεί να είναι 300 ε, ή οτιδήποτε άλλο ευρώ ή οτιδήποτε, πάντως ξεπερνάει αυτό. Γι' αυτό θα ήθελα να ζητήσω σε αυτές τις περιπτώσεις που επαναλαμβάνονται πάρα πολλές φορές για πολλούς από εμά να υπάρξει μια πιο εκπεφρασμένη ρύθμιση ώστε να μην είμαστε υποχρεωμένοι κάθε φορά όταν πρέπει να διανεκτερεύσουμε κάπου λόγω μιας ε, εκδήλωσης την οποία δεν μπορούμε να αποφύγουμε να ζητήσουμε και πάλι η Συμβουλευτική Επιτροπή να γνωμοδοτήσει για το αν αυτή η εκδήλωση ήταν κατά τα 100% μέσα στα πλαίσια της εντολής μας ως ευρωβουλευτές ή όχι. Και για την τροπολογία 9, <clears throat> για τα έσοδα τα οποία ε, αποκτά κανείς, νομίζω ότι είναι σημαντικό να μπορεί κανείς να δίνει κάποιες εξηγήσεις για τα θέματα αυτά. Σε ορισμένε περιπτώσεις στη Γερμανία, όταν είναι ε, παντρεμένος κάποιος ε, ε, βουλευτής, αν κάποιος είναι παραδείγματος χάρη γε, γεωργός, θα πρέπει θεωρητικά να δηλώσει και το εισόδημα της συζύγου του μαζί με το δικό του. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα μέσα στο σύστημα δήλωση εισοδημάτων να έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε μικρές παρατηρήσεις και να εξηγήσουμε ότι μπορεί να έχει προκύψει μια τέτοια ε, περίπτωση και καταλογίζεται και το εισόδημα κάποιου άλλου ατόμου μαζί με το δικό του. Επίσης υπάρχουν και δραστηριότητες τις οποίες εγώ έχω ασκήσει στο παρελθόν από τις οποίες μπορεί ακόμα να παίρνω κάποια χρήματα. Θα ήθελα λοιπόν να έχω το, τη δυνατότητα μέσα στη δήλωση να κάνω κάποια επεξήγηση που να λένε ότι αυτές είναι, αυτά είναι χρήματα τα οποία έρχονται από δραστηριότητε που ίσχυσα σε τοπικό επίπεδο ως βουλευτής στο παρελθόν. Αυτό νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο είναι απαραίτητο για να μπορεί να αποφύγουμε καταστάσεις όπου θα μας βγάζουν στις εφημερίδες και θα λένε ότι ο τάδε βουλευτής βγάζει πέραν του μισθού του και τόσα περαιτέρω ποσά όταν δεν έχει πια κάποια άλλη δραστηριότητα εκτός του Κοινοβουλίου. Αυτά τα σημεία λοιπόν νομίζω ότι αξίζει να τύχουν κάποιες διευκρίνησεις. Ευχαριστώ. Ο Μέντες Δεβίγο για μια προσθήκη σύντομα και ο συνάδελφος Γκρέτε. Και ακόμη ένας. Εγώ θα είμαι πολύ σύντομος. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Βέσσερ Σμίτη για την παρέμβασή του. Έχει πολύ δίκιο. Σε μία αναθεώρηση του κανονισμού δεν μπορούμε να τροποποιήσουμε το πρωτόκολλο των ασυλιών. Είναι αδύνατον. Εμένα θα μου άρεσε να, μέσα από τον κανονισμό να αλλάξω και το εκλογικό σύστημα και το πρωτόκολλο των ασυλιών. Ο κύριος Μέσερ εισηγείται μία αλλαγή. Αν ο κύριος Μέσερ υποβάλει μία αίτηση για αλλαγή των ασυλιών και του εκλογικού συστήματος θα τον υποστηρίξουμε. Κύριος Γκρότ. Μία ερώτηση για τους εισηγητές. Πόσο συχνά έχει παρουσιαστεί στο παρελθόν ένας εισηγητής να, αποσυρθεί, να του αποσυρθεί η έκθεση ναι. ή να την αποσύρει μόνος του λόγω δυσκολιών. Γιατί το συζητάμε και θα ήθελα να ξέρω πόσες συγκεκριμένες περιπτώσεις έχουν υπάρξει κατά το παρελθόν. Τι πράγμα συζητάμε δηλαδή για τη διαμόρφωση του μηχανισμού κυρώσεων. Ίσως θα μπορούσατε να απαντήσετε στην ερώτηση αυτή. Ίσως να είναι και πολύ περίπλοκο και να μην έχετε κάποια έτοιμη απάντηση. Ο κύριος Σόντεργαρτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πάρα πολύ σύντομα για τον κύριο Χέφνερ. Εγώ δεν θέλω εδώ να ξεκινήσω μία συζήτηση περί κομμουνισμού με τον κύριο Χέφνερ. Δεν έχω ετοιμάσει κάτι τέτοιο. Θα ήθελα απλώς να πω κάτι. Αυτό για το οποίο μιλάμε εδώ σήμερα είναι το εξής. Εμείς το καθιστούμε μία υποχρέωση εξυπηρέτησης του, του γενικού συμφέροντος δεσμευόμαστε να υπερασπιστούμε το γενικό συμφέρον. Δεν μπορούμε εμείς να επαληθεύσουμε αν πληρείται ή όχι το γενικό συμφέρον. Οι στόχοι των πρασίνων είναι πολύ πιο ε, σημαντικοί από ότι η βιομηχανική επιβίωση. αλλά ε, η επιβίωση της βιομηχανίας αποτελεί καθολικό συμφέρον, δεν ξέρω, ε, είναι πράγματα τα οποία δεν, δεν ορίζονται, δεν υπάρχουν ορισμοί γι' αυτό. Πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί. Τι θέλει να πει κάτι, ποιο είναι το νόημα. Φυσικά και είμαστε υποκειμενικοί όταν προχωράμε σε μια τέτοια προσέγγιση, σύμφωνη αλλά πρόκειται για λόγια κενά περιεχομένου, τα οποία δεν λένε τίποτα στον κοσμάκι μια σύντομη παρατήρηση. Η πολιτική σημαίνει να εργάζεται κανείς για το γενικό καλό. Και όλες αυτές οι κυρώσεις οι οποίες αναφέρονται εδώ πέρα ε, δεν παρεμβαίνουν όταν πει κάποιο ότι ο κ. Σόντεργαρντ και ο κ. Χέφνερ δεν υπηρετούν το κοινό καλό, αλλά όταν έχουν διαπράξει μια συγκεκριμένη πράξη, η οποία παραβιάζει του κανόνε. Ωραία. Λοιπόν, αντιδρώ κι εγώ και θα πω τη γνώμη μου για όλη αυτή τη συζήτηση, ήταν πολύ πλούσια. Κάποιος από εσά είπε, που δεν θυμάμαι ποιος ήταν, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί, ό,τι περνά από τα χέρια του για να έχει την εμπιστοσύνη των εκλογέων. Αυτό σημαίνει τι, σημαίνει διαφάνεια, αυστηρούς κανόνες, αρκετά αυστηρούς κανόνες, για τη συμπεριφορά των ε, διαφόρων βουλευτών. Αυτό συνοδεύεται, αυτό ε, επιβεβαιώνει και την πρόθεσή μας να καταλήξουμε να καταλήξουμε στην διόρθωση του κώδικα διοντολογία. Γιατί όμω ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία έτσι στα γρήγορα. Διότι διαπιστώσαμε ότι υπήρχαν τρεις περιπτώσεις ε, ε, πρόβλημα ε, διαφθοράς. Αυτό θα το αποφασίσουν βέβαια οι δικαστέ, αν, αν υπάρχει όντω αδίκημα. Πάντως ξεσηκωθήκαμε και είπαμε τέρμα εδώ σε αυτό το κοινοβούλιο θέλουμε διαφάνεια. Υπάρχει αυτό λοιπόν ο κώδικα, σε αυτόν τον κώδικα διοντολογία υπάρχει Είπα... Ε, ε, και ε, υπησέρχεται μάλλον η έννοια του κηρύγματος. Θέλουμε να αντιδράσουμε και να διακηρύξουμε γρήγορα. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να αποφασίσουμε γρήγορα. Και ζητούμε και από τα εθνικά κοινοβούλια. Πρόκειται για έναν κώδικα δεοντολογίας αυτός ο κώδικας ιδεοντολογίας να βρίσκεται υπεράνω των κωδίκων δεοντολογίας των Εθνικών Κοινοβουλίων. Θέλουμε να αφήσουμε κατά μέρο ε, τις δευτερεύουσες διορθώσεις και να στοχεύσουμε μόνο στα ουσιαστικά. Εγώ τα σημείωσα όλα όσα που μου είπατε, μερικά από αυτά που μου είπατε φυσικά πρέπει να τα ξανασκεφτώ. Δεν μπορώ ευθύ αμέσω να πω τη γνώμη μου, αλλά μερικά πράγματα μπορώ να σας τα απαντήσω. Σας ανέφερα ήδη την ε, διαφορά μεταξύ του εκλογικού αξιώματος που αναθέτει ο λαός και του εκλογικού αξιώματος ε, που αναθέτει η Ολομέλεια. Εγώ κατάλαβα ότι για την άρση του ορισμού ως εισηγητή είναι η αρμόδια επιτροπή αυτή που μπορεί να την εγκρίνει. Εγώ κατάλαβα ότι αυτή η κύρωση που δεν προβλέπεται από το άρθρο 153 ε, εισάγεται χωρίς όμως να βρίσκεται στο τέλος γιατί η τελευταία κύρωση είναι η ανάκληση του εκλογικού αξιώματος. Για το εκλογικό αξίωμα και την ανάκληση του αποφασίζει η διάσκεψη των Προέδρων με τα δύο τρίτα και μετά η Ολομέλεια και η Ολομέλεια ε, επικυρώνει αυτή την ε, κύρωση με τα δύο τρίτα πάλι των ψήφων και αυτό για να αποπολιτικοποιήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο την υπόθεση. Η τέταρτη κύρωση που προβλέπεται από την ομάδα εργασίας, η τέταρτη πια είναι αλήθεια, ψάχνει ο πρόεδρος, προβλέπει ότι σε περίπτωση παραβίασης του κώδικα δεοντολογίας από έναν εισηγητή κατά την άσκηση των καθηκόντων του ως εισηγητή μπορεί να θέσει ο πρόεδρος της Επιτροπής το ζήτημα στη διάσκεψη των προέδρων. Γιατί όμως αυτό το σημείο 4 δεν λέμε το ίδιο πράγμα που λέει και το σημείο 5 ότι η διάσκεψη των Προέδρων μπορεί να εφαρμόζει το άρθρο 19 οπότε ζητά από την Ολομέλεια να το εφαρμόσει. Εδώ υπάρχει σιωπή γύρω από το, γύρω από το θέμα. Μου φαίνεται να κατάλαβα ότι ο η θέση που βγαίνει από εδώ ως επικρατέστερη είναι ότι η αρμόδια επιτροπή είναι αυτή που μπορεί να ανακαλέσει. Εγώ όμως τονίζω το εξής. Το in senso proprio, cioè per nomina dovuta all'Assemblea, Presidente, Vicepresidenti, Questori, eccetera. Ρωτώ εγώ. Για την ανάκληση του αξιώματος το σώμα αποφασίζει στα δύο τρίτα. Στην Επιτροπή όταν πρέπει να ανακαλέσουμε τον ορισμό σε εισήγηση θα πρέπει να έχουμε πάντα την ίδια αναλογία των δύο τρίτων. Σας το ρωτάω εγώ αυτό και εσείς σκεφτείτε το. Μπορείτε βέβαια να καταθέσετε ό,τι τροπολογία θέλετε και έχουμε χρόνο για να το σκεφτούμε παραπάνω. Να πω όμως και κάτι άλλο για το θέμα της ε, Συμβουλευτικής Επιτροπής. Μα πρόκειται για Συμβουλευτική Επιτροπή. Δεν συμβουλεύει, ε, δεν αποφασίζει, συμβουλεύει. Και η γνώμη δεν είναι δεσμευτική. Σίγουρα υπάρχει κάποιο διαδικαστικό πρόβλημα που θα προκύψει και όπως είπε και ο κύριος Ντάφ. Το κείμενο το οποίο πρότεινα εγώ είναι το κείμενο της ομάδας εργασίας και προβλέπει ότι ο ενεχόμενος ε, βουλευτής ε, θα πρέπει να εισακουστεί από τον πρόεδρο. Αυτή η διαδικασία προβλέπεται και για την Επιτροπή, Συμβουλευτική Επιτροπή. αυτή η συμβουλευτική επιτροπή θα μπορούσε να συντάξει έναν κανονισμό και μετά αυτός ο κανονισμός να εγκριθεί από τον πρόεδρο αλλά στην τελευταία τροπολογία που εγώ πρότεινα και που ανταποκρίνεται και στο κείμενο της ομάδας εργασίας είναι η τροπολογία 14 και που λέει ότι Η Συμβουλευτική Επιτροπή μπορεί να προτείνει τροποποίηση του κώδικα δεοντολογίας, ε, να αναθεωρήσει τις ποινές κλπ. Θα μπορούσε κάλλιστα λοιπόν να αναλάβει και την επεξεργασία ενός κανονισμού για την Συμβουλευτική, η Συμβουλευτική Επιτροπή. Για το άρθρο 1, συνάδελφε Σόντεργαρτ, η ομάδα εργασίας είχε ετοιμάσει ένα νέο κείμενο το οποίο ονόμαζε «Γενικές Αρχές». Εμένα μου φάνηκε ότι στην απαρίθμηση των τεσσάρων σημείων μετά τον τίτλο δύο έχουν ενδεικτικό χαρακτήρα. Λέει ότι θα πρέπει να συμπεριφέρεται ο βουλευτής με ανιδιοτέλεια, κεραιότητα, διαφάνεια, και τι ημιότητα μπορεί να μην αρέσουν οι όροι. Εντάξει, σίγουρα δεν διαπιστώνουμε συγκεκριμένα τους... Ε, δεν μπορούμε να διαπιστώνουμε σε συγκεκριμένες καταστάσεις όλες αυτές τις συμπεριφορές. Αλλά το Γ και το Δ αναφέρουν όμως ότι οι βουλευτές δεν θα πρέπει να δέχονται δωρεές ή δώρα σε είδος. Δηλαδή εκεί πλέον έχουμε συγκεκριμένη παραβίαση. Εσείς κάλλιστα μπορείτε να ασκήσετε κριτική και να υποβάλλετε τροπολογίες. Εγώ πιστεύω πάντως από άποψη ορολογίας να διακάνουμε διάκριση μεταξύ των αρχών και των υποχρεώσεων. Τώρα εγώ δεν ξέρω αν υπήρχαν προηγουμένως ε, ε, ποινές ανάκλησης ε, δεν νομίζω γιατί δεν ε, προβλεπόταν η ανάκληση ως ποινή στην παραβίαση του κώδικα διοντολογίας. Για το θέμα των Intergroup. Πράγματι όπως λέει ο συνάδελφος Μέντες και σήμερα υπάρχει ο κανόνας ότι κάποιος θα πρέπει να δηλώνει το λέμε στον τωρινό κώδικα διοντολογίας. Αλλά το είχαμε ξεχάσει αυτό το κείμενο. Πιστεύω, όπως είπε και ο κύριος ε, Μέντες, ε, θα πρέπει να υπεραμυνθούμε αυτού του κειμένου. Επειδή αποκλείεται να μιλήσουμε γι' αυτό στις ε, αρχικές διακηρύξεις, τότε θα πρέπει να μιλήσουμε για τα intergroup χωριστά. Συνάδελφε Μπρο, λέτε ότι το ένα της τροπολογίας εννιά σας φαίνεται πολύ γενικό. Μα. Ότι θα πρέπει να δηλώνουν οποιοδήποτε οικονομικό συμφέρον το οποίο μπορεί να ε, επηρεάσει της ε, την άσκηση των ε, βουλευτικών καθηκόντων. Ε, μα ξέρετε όμως πρόκειται για ένα εδάφιο συμπερασμάτων, οπότε είναι που ο νομοθέτης φοβάται και το ξαναβάζει και το βάζει γενικά. Τώρα για για την ανάκληση από τον πρόεδρο. Εμείς ε, θέλουμε την αποπολιτικοποίηση στο θέμα δηλαδή της ανάκλησης και θέλουμε να είμαστε υπεράνω των μερών. Ο πρόεδρος είναι Uber Είναι υπεράνω όλων των πολιτικών παρατάξεων. Τώρα, όταν μεσολάβησαν όλα αυτά τα επεισόδια τα οποία πραγματικά επιτάχυναν τη διαδικασία επεξεργασίας του κώδικα διοντολογίας, Διαπίστωσα ότι εμείς τι κάνουμε, προσπαθούμε να εγγυηθούμε την ακαιρεότητα των βουλευτών και τιμωρούμε αυτούς οι οποίοι υπόκεινται στο αντίκημα της δωροδοκίας. Αλλά μετά ποιος τους τιμωρεί. Αλλά στη συνθήκη της Λισαβόνας, την οποία θα πρέπει να ξαναπάρουμε στα χέρια μας, να τη διαβάσουμε και να την ξανασκεφτούμε, μόνο υποθεσμικού προφίλ βέβαια, αυτή η δυνατότητα που μας δίνεται στο άρθρο 86 να έχουμε έναν Ευρωπαίο εισαγγελέα ο οποίος θα πρέπει να ασχολείται με την έρευνα και την άσκηση της ποινική δράσης για οικονομικά δικήματα κατά της Ένωσης. Στην τελευταία παράγραφο του άρθρου 86 προβλέπει ότι αυτός ο εισαγγελέας μπορεί να έχει αρμοδιότητα και για όλα τα σοβαρά διασυνοριακά αδικήματα. Βέβαια θα μου πείτε ε, εκεί έχουμε την εθνική κυριαρχία, το ποινικό δίκαιο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα κράτη-μέλη. Αλλά αν εμείς δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε διερευνητικές διαδικασίες και ανακρίσεις για αυτού του είδους ε, τα αδικήματα ε, νομίζω ότι αυτό πρέπει να το καλύψουμε διότι σήμερα έχουμε στη συνεργασία στα πλαίσια του Σέγγεν θα έπρεπε να αρχίσουμε να το σκεφτόμαστε το θέμα να γίνεται να εκτελήσεται η ανακριτική διαδικασία και μετά να πηγαίνει σε εθνικό επίπεδο εγώ δεν ξέρω τι έγινε με αυτούς τους τρεις δημοσιογράφους που ήρθαν εδώ στο κοινοβούλιο και προσπάθησαν να διαφθείρουν ε, τους ε, βουλευτές ως τι θα καταδικαστούν και ως ε, προβοκάτορες, ως διαφθορείς, ως δωροδοκητές, σαν τι. Αυτό εξαρτάται από τα κράτη-μέλη. Ξέρετε, εγώ επιβίωσα από, ένα πρόσφατο, ε, από μια πρόσφατη συνάντηση στο Παρίσι με εισαγγελείς για τη δημιουργία του Ευρωπαίου εισαγγελέα και πρέπει να το σκεφτούμε. Τώρα, έχουμε την προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών και αν θέλουμε να ολοκληρώνουμε γρήγορα τις εργασίες μας θα πρέπει να ορίσουμε ως προθεσμία την 27η Οκτωβρίου στις 9 το πρωί για να μπορέσουμε μετά να ψηφίσουμε σε μία έκτακτη συνεδρίαση στις 14 Νοεμβρίου στο Στρασβούργο. Εάν συμφωνείτε, ούτως ε, αποφασίζουμε. Πάμε τώρα στο επόμενο θέμα που είναι, ε, πρόκειται για την πρωτοβουλία πολιτών. Στην προηγούμενη συνεδρίαση των συντονιστών εξετάσαμε δύο δυνατότητες σχετικά. Πώς να προετοιμαστούμε για, την, ε, για αυτήν την πρωτοβουλία πολιτών που θα καταστεί λειτουργική την 1η Απριλίου του 2012. Ο κύριος Χέφνερ ζήτησε η Επιτροπή μας να συντάξει μία έκθεση πρωτοβουλίας Η κυρία Γκουρμάη έχει και μία επιστολή του κυρίου Ραμασούρ που λέει ότι θα πρέπει να προετοιμάσουμε την μεταρρύθμιση ή την τροποποίηση του κανονισμού. Η κυρία Γκουρμάη έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε φυσικά ποιος είναι ο σκοπός της συζήτησης αυτής. Να δούμε πώς θα εφαρμοστεί η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία και ο σχετικός κανονισμός ε, του Κοινοβουλίου και φυσικά να αποφασίσουμε ποια θα είναι η καλύτερη διαδικασία να γίνει η εφαρμογή αυτή. Όπως ανέφερε και ο πρόεδρος Καζίνη, ο κύριος Λαμασούρ δεν μπορεί να παρευρεθεί εδώ γιατί προεδρεύει τις ε, συνεδρίες της Επιτροπής Προϋπολογισμού αλλά, όπως τα ξέρετε, ο κανονισμός για την Ευρωπαϊκή αυτή πρωτοβουλία προβλέπει την διεξαγωγή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημόσιας ακρόασης σε περίπτωση που συγκεντρωθούν ένα εκατομμύριο υπογραφές και ασφαλώς ελπίζουμε αυτό να παρουσιαστεί σε πολλές περιπτώσεις. Και χαίρομαι που η Επιτροπή και το Συμβούλιο παρευρίσκονται εδώ, γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η κοινή εργασία. Πρώτα, πήγε κάτι εντελώ καινούριο. και προφανώς θα πρέπει να γίνουν κάποιοι τροποποιήσεις στον κανονισμό του Κοινοβουλίου σχετικά με αυτό. Και φυσικά ο Άλαν Λαμασούρ και εγώ είχαμε καταρχάς υπόψη και σκεφτόμαστε το θέμα αυτό εδώ και καιρό σε ό,τι αφορά τη μορφή των απαραίτητων αυτών αλλαγών. Τι σκοπεύουμε να κάνουμε εύκολη, άμεση και γρήγορη διαδικασία γιατί τον Απρίλιο του 2012 θα τη εφαρμογή ο κανονισμός αυτός. Θέλουμε λοιπόν να προτείνουμε κάποιες αλλαγές ε, στον κανονισμό βάσει του άρθρου 212. Δεν είναι δύσκολο το εγχείρημα. Είμαστε ήδη έτοιμοι. Και φυσικά στο πνεύμα της καλής συνεργασίας θα θέλαμε όλα αυτά να υπογραφούν και με τον κύριο Χέφνερ και με την Ταϊάννα να σας υπενθυμίσω ότι η Επιτροπή Αναφορών έκανε πολύ σημαντική δουλειά μαζί μας επί αυτής της σημαντικής έκθεσης. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη τώρα? Ότι όταν αυτά υποβληθούν στον πρόεδρο Μπούζεκ θα επανέλθουν στην Επιτροπή μας καθότι είμαστε υπεύθυνοι για τον κοινωνισμό και θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε ενδεχόμενες τροπολογίες. Μετά θα εγκριθεί, θα περάσει στην Ολομέλεια για επίσημη έγκριση, προκειμένου να ενταχθεί στο σώμα του κανονισμού. Είμαστε πεπισμένοι ότι έτσι θα υπάρχει ευκαιρία για συζήτηση στην Επιτροπή και έτσι θα διασφαλιστεί ότι θα είμαστε έτοιμοι πριν τον Απρίλιο. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί φίλοι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ασφαλώς ε, πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην διαδικασία της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας. Να μην ξεχνάμε όμως ότι η πρωτοβουλία αυτή των Ευρωπαίων πολιτών αφορά βασικά τους πολίτες και όχι τους βουλευτές. Αυτόν το θυμόμαστε στην όλη συζήτηση. Μία έκθεση πρωτοβουλία ίσω να ε, υπογράμμιζε υπερβολικά το ρόλο του Κοινοβουλίου και να δημιουργούσε φρούτε ελπίδε. Δεν θέλουμε να δώσουμε την εντύπωση ότι μπορούμε να επηρεάσουμε εμεί στο Κοινοβούλιο την απόφαση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλουμε να βρούμε ένα πρακτικό τρόπο μόνο να διοργανωθεί η ακροασία. Να είμαστε λοιπόν ακριβεί και συγκεκριμένοι. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει ασφαλώς ε, μέσω πολλών νομοθεμετημάτων την ε, πρωτοβουλία των Ευρωπαίων πολιτών. Είναι όλα αυτά τόσο καταφανή που δεν βλέπουμε την ανάγκη να υπάρχει, ανάγκη μάλλον για μια ε, έκθεση πρωτοβουλίας. Έχουμε λοιπόν πολλές ε, δυνατότητε και δεν είναι καλό να αυτοπεριοριζόμαστε σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο των προτινόμενων αλλαγών. Έχουμε κάποιες σκέψεις με τον κύριο Λαμασούρ. Η ακρόαση αυτή θα πρέπει να διοργανώνεται από την καθήλυν αρμόδια Επιτροπή, να συνεργάζονται και οι συναρμόδιες επιτροπές. Η διάσκεψη των Προέδρων θα πρέπει να αποφασίζει κατά περίπτωση ποια θα είναι η καθήλυνα αρμόδια επιτροπή και η ακρόαση θα πρέπει να διεξάγεται εντός τριών μηνών από την έναρξη και την κατάθεση της πρωτοβουλίας ενώπιον της Επιτροπής και προτού η Επιτροπή παρουσιάσει τα αποτελέσματά της, τα συμπεράσματά της. και ε, σε περίπτωση που γίνει αποδεκτή η πρωτοβουλία θα περάσει στην ατζέντα αυτόματα της διάσκεψης των Προέδρων. Η αναγνώριση της ε, εμπειρίας της Επιτροπής ε, Αναφορών στην αντιμετώπιση τέτοιων πολιτών σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθούν τα 1 εκατομμύριο υπογραφών αλλά υπάρχει πολιτική ανάγκη, θεωρούμε ότι είναι κάτι σημαντικό επίσης. Μπορούμε λοιπόν να προτείνουμε και μία εναλλακτική τέτοια οδό. Η λύση αυτή θα δώσει και μία εγγύηση για τους διοργανωτές της συλλογής υπογραφών, γιατί ξέρετε πόσο δύσκολο ή εύκολο μπορεί να είναι το έργο αυτό. Αυτό λοιπόν είναι κάτι στο οποίο θα πρέπει να επιδείξουμε ιδιαίτερη προσοχή γιατί σημαίνει μεγάλο όγκο εργασία για τους πολίτες και θα πρέπει να υπάρχουν κατά κάποιο τρόπο κίνητρα. Αν θα μπορούσατε λοιπόν να μου γνωστοποιήσετε την γνώμη σας για όλα αυτά. Αλλά το πολύ σημαντικό είναι να έχουμε κάτι έτοιμο μέχρι τον Απρίλιο. Ο συνάδελφος ε, Χέφνερ και μετά ο συνάδελφος Σόμπλερ. Αγαπητοί συνάδελφοι, έκανα την πρόταση αυτή για μια έκθεση πρωτοβουλίας πριν από μήνες ήδη, πριν τις θερινές διακοπές, γιατί πολύ απλά πιστεύω ότι είναι σημαντικό το έργο που έχουμε να επιτελέσουμε εδώ. Αυτό το μωρό, αν θέλετε, αυτό το παιδί, το δημιούργημά μας, θα πρέπει να του δώσουμε την ανάλογη προσοχή, προκειμένου να αναπτυχθεί σωστά και να λάβει μια σωστή μορφή. Συνολικά θα πρέπει να πούμε ότι ο κανονισμός για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών ήταν μεγάλη επιτυχία. Το Κοινοβούλιο κατάφερε να εισάγει και πολλά δικά του σημεία, τα οποία θεωρώ ότι βελτίωσαν περαιτέρω την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παρόλα αυτά εξακολουθεί να είναι απόλυτα ανοιχτό κατά πόσο θα στεφτεί με πραγματική επιτυχία το εγχείρημα ή όχι. Και νομίζω ότι αυτό θα εξαρτηθεί από το πώ θα διαμορφωθεί ε, στην πράξη η διαδικασία. Ιδιαίτερα η διαδικασία στο εσωτερικό του Κοινοβουλίου αλλά και μεταξύ Επιτροπής Κοινοβουλίου και Πολιτών. Αυτό είναι που δεν ορίζεται στον κανονισμό. Άρα μιλήσαμε και ορίσαμε με μεγάλη λεπτομέρεια το πώς θα συλλέγονται οι υπογραφές, από ποιες χώρες, πώς θα γίνονται οι υπολογισμοί, με βάση ποιους πίνακες, πώς θα ελέγχονται οι υπογραφές. Αλλά δεν είπαμε τίποτα, δεν ρυθμίσαμε τίποτα για το τι θα συμβεί μετά και το πώς θα διοργανωθεί η μετέπειτα διαδικασία. Και αυτό νομίζω ότι ε, μας κάνει να σκεφτόμαστε πολλά θέματα τα οποία δεν έχουν απαντηθεί επαρκώς. Και θεωρώ ότι πολλά ερωτήματα δεν αφορούν μόνο εμάς ως Κοινοβούλιο, αλλά και διαθεσμικά ζητήματα σε ό,τι αφορά τις σχέσεις Κοινοβουλίου και Επιτροπής. Να πω επί της αρχής ότι το όλο όργανο, το, το όλο εργαλείο δεν αποτελεί ένα εργαλείο της άμεσης δημοκρατίας, δημοκρατίας αποφάσεων. Πρόκειται για συμμετοχική δημοκρατία. Αν καταφέρουμε να το διαμορφώσουμε με θετικό τρόπο, πρέπει να υπάρχει διάλογος, να υπάρχει διάλογος μεταξύ των πολιτών και των θεσμικών οργάνων, να δοθεί εντύπωση στους ε, πολίτες ότι τα συμφέροντά τους θα εισακούν τα θεσμικά όργανα. Δεν μπορούμε να υποσχεθούμε κάτι παραπάνω. Δεν μπορούμε να υποσχεθούμε στους πολίτες ότι αν ε, συλλέξουν ένα εκατομμύριο υπογραφές για ένα σκοπό θα πραγματοποιηθεί ο σκοπός αυτός. Δεν είναι αυτός ο σκοπός της πρωτοβουλίας. Γι' αυτό λοιπόν όλα εξαρτώνται από το πώς θα διοργανωθεί αυτή η διαδικασία, πώς θα γίνουν αυτές οι επαφές. Αν έχουμε δύο τρένα, το ένα δίπλα άλλο, τους ε, πολίτες που συλλέγουν τις υπογραφές και κάνουν τα θεσμικά όργανα τη δουλειά τους, αλλά αν κινούνται παράλληλα χωρίς να συναντηθούν ή κινηθούν προς διαφορετικές κατευθύνσεις που με ανησυχεί ιδιαίτερα γιατί αυτές οι διαδικασίες μπορούν να κινηθούν προς διαφορετική κατεύθυνση και αυτό με ανησυχεί πραγματικά. Αυτό δεν θα ενδυναμώσει θα αποδυναμώσει μάλλον τη δημοκρατία. Το θέμα λοιπόν είναι πώς ε, θα μπορέσουμε αυτές οι τροχές να μην είναι παράλληλες, αλλά πώς μπορούν να συνενωθούν τα δύο τρένα αυτές, τα δύο τρένα αυτά, προκειμένου οι εργασίες του Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εκεί βρίσκεται, αν θέλετε, η δυσκολία να μην προκύψουν ατυχήματα. Και σας το λέω αυτό μετά από μεγάλη εμπειρία, 36 χρόνια σε ό,τι αφορά την συμμετοχική δημοκρατία σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πολύ δύσκολο να μην απογοητευτεί ο κόσμος, ούτε και εμείς όμως να υποσχεθούμε κάτι το οποίο δεν μπορούμε να πραγματοποιήσουμε. Θα πρέπει λοιπόν ο πολίτης να αισθανθεί ότι εισακούεται, αλλά και εμείς να είμαστε απόλυτα ελεύθεροι στις ενέργειές μας, προκειμένου να μην πιεστούμε στη λήψη αποφάσεων. Και γι' αυτό λοιπόν πολλά σημεία θα πρέπει να κοιτάξουμε. Στο τι θα συμβεί για παράδειγμα αν ε, συλλεχθούν ένα εκατομμύριο υπογραφές και ε, είναι όντως αποδεκτό και παραδεκτό το αίτημα. Ο κανονισμό ορίζει αυτή την ιδέα των ακροάσεων, αλλά ήταν μέχρι τελευταία στιγμή αμφιλεγόμενο το θέμα αυτό. Τελευταία στιγμή λοιπόν βρήκαμε, πραγματικά την τελευταία στιγμή, βρήκαμε στον τρομερή διάλογο ένα συμβιβασμό και είπαμε ότι υπάρχει ε, αξίωση για, τέτοιο, για μια τέτοια ακρόαση και είπαμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διασφαλίσουν διεξαγωγή ακρόασης ε, και θα υπάρχει αντιπροσώπευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, κατά περίπτωση. Σκοπός είναι να διασφαλιστούν λοιπόν όλα αυτά, αλλά θα πρέπει να διευκρινιστεί το κατά πόσον, για παράδειγμα, πώς θα ελέγξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το αίτημα και πώς θα ενημερώσει το Συμβούλιο. Ποιος είναι υπεύθυνο στο Κοινοβούλιο για να κάνει τις διαπραγματεύσεις με το Κοινοβούλιο για την διεξαγωγή της ακρόασης προκειμένου να τηρείται το χρονοδιάγραμμα και του Κοινοβούλιου και της Επιτροπής. Ποιος θα εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει όλα αυτά να μην τα ρυθμίσουμε μόνο εμείς στο Κοινοβούλιο, να τα συμφωνήσουμε και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να λειτουργήσουν στην πράξη. Ποιο θα συμμετάσχει λοιπόν, ποιο θα εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τι χρονικό περιθώριο θα πρέπει να δοθεί σε μια τέτοια ακρόαση γιατί σε πολλές ε, συνομιλίες έχω ακούσει πάρα πολλές διαφορετικές ε, προθεσμίες. Ποιο, τι μορφή θα έχει αυτή η ακρόαση φτάνει η Επιτροπή Αναφορών, θεωρώ πως όχι, αλλά αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί. Μήπως χρειάζεται ένα ειδικό όργανο, μήπως θα είναι κάποια εξειδικευμένη επιτροπή μαζί με την Επιτροπή Αναφορών, ποιος θα είναι ο ρόλος ε, των επιτροπών αυτών, ποιος θα έχει ποια δικαιώματα, ποιος θα έχει δικαίωμα απόφασης, πόσους πολίτες θα καλέσουμε, τι κόστος επιτρέπεται, ποιο κόστος καλύπτεται, ποιο κόστος δεν καλύπτεται. Ξέρετε ότι εμένα τα θέματα αυτά με απασχολούν εδώ και πάρα πολύ καιρό και το έχω κάνει αυτά σε διάφορες χώρες και ξέρω ποια είναι τα ερωτήματα που ανακύπτουν. Εγώ λοιπόν πρότεινα να καταρτιστεί μία έκθεση πρωτοβουλία, γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι ο κατάλληλος τρόπος εργασίας να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Η έκθεση πρωτοβουλίας επίσης θα πρέπει να περιλαμβάνει και μια, ένα αίτημα αλλαγή του κανονισμού. Αλλά αυτό θα το ρυθμίσουμε. Θα ήθελα αυτό να γίνει με τέτοιο τρόπο προκειμένου όσοι ασχολούνται με το θέμα αυτό, ήταν αναγόλες ο, ο Αλάν Λαμασούρ και η κυρία Ζερμάη, να μπορέσουν να συζητήσουν τα θέματα αυτά αλλά θα πρέπει όλα αυτά να γίνουν με τρόπο που να ρυθμίζει όλα αυτά τα θέματα, να τα διευκρινίζει και να μην αφήνει ανοιχτά βασικά ζητήματα. Γιατί από την εμπειρία μου να σας πω ότι όποτε μένουν ανοιχτά τέτοια θέματα, για τον κανονισμό για παράδειγμα, αν δεν ρυθμίσουμε πια επιτροπή, ότι ο πρόεδρος της Επιτροπής αποφασίζει, η διάσκεψη των προέδρων αποφασίζει σε ό,τι αφορά το κόστος, την κάλυψη του κόστους. Α, όλα αυτά δεν θα πρέπει να μείνουν ανοιχτά γιατί θα προκαλέσουν ε, καυγάτες, που δεν χρειαζόμαστε. Θα πρέπει μέσα από τον κανονισμό λοιπόν να ικανοποιούμε τους πολίτες. Γιατί ξέρετε, η ίδια η πρωτοβουλία είναι η συμμετοχική δημοκρατία. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την επιτυχία ενός τέτοιου αιτήματο της πρωτοβουλίας των πολιτών. Όλα αυτά λοιπόν που έχουν μείνει ε, ανοιχτά θα πρέπει να τα ρυθμίσουμε. Ο Σέπλιν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Γοντεμάιο. Μιλώ εξ ονόματος του ΕΛΚ γιατί ο κύριος Μέντες Δεβίγο αναγκάστηκε να φύγει και μα έχει δώσει μια πολύ σωστή παρουσίαση για το πώ έχει η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Εμεί υποστηρίζουμε γενικά αυτή τη διαδικασία εν γέννη με κάθε σεβασμό στον κύριο Χέφνερ δεν υποστηρίζουμε μια έκθεση πρωτοβουλία σε αυτό το στάδιο. Νομίζω ότι τα περισσότερα στοιχεία υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Το νέο αυτό λοιπόν εργαλείο, η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών μπορεί να είναι μια επιτυχία και οι διαδικασίες που έχουμε αυτή τη στιγμή μπορούν να ξεπεράσουν όλες τις αμφισημίες. Πάντα θα υπάρχουν ένα Έτσι είναι η ζωή. Αλλά όλα αυτά μπορούν πραγματιστικά και στην πράξη να ξεπεραστούν. Εγώ συμφωνώ ότι μιλάμε εδώ για μία συμμετοχική δημοκρατία και διάλογο πολιτών και θεσμικών οργάνων. Αλλά δεν πρέπει να ακολουθήσουμε το δρόμο της υπερβολικής ρύθμισης. Η υπερβολική ρύθμιση πάντα δημιουργεί μια κατάσταση στατικότητας, ε, εμποδίζει την πραγματική αποτελεσματικότητα αυτών των εργαλείων. Και αν έχουμε παγιωμένους κανόνες οι οποίοι ούτως ή άλλως θα δημιουργηθούν. Όλα αυτά απαιτούν ερμηνεία, δημιουργούν περαιτέρω αμφιβολίες και αμφισημίες. Δεν νομίζω ότι προς το παρόν αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό. Ίσως θέλουμε περισσότερη ευελιξία και όχι το αντίθετο. Κύριε Χεύνα, ίσως έχουμε και μια σύγκρουση πολιτιστικού χαρακτήρα. Κάποιες κουλτούρες θέλουν πιο σαφείς ρυθμίσεις από ό,τι, όλες οι, από ό,τι άλλες. Ίσως εκεί είναι η διαφωνία μας. Ο κύριος Γκερέρο πρέπει να μιλήσει και πάλι. Ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ σύντομα. Όταν ξεκινήσαμε όλη αυτή την ε, δουλειά για την οργάνωση της ε, πρωτοβουλίας ε, πολιτών, ξέραμε ότι έπρεπε να το κάνουμε γρήγορα, διότι εντασσόταν αυτή η πρωτοβουλία μέσα στη συνθήκη της Λισαβόνας που απευθυνόταν κατευθείαν στους πολίτες και ήταν σαφές ότι θα έπρεπε να λειτουργήσει κατά την πρώτη χρονιά ή στο τέλος της ε, ε, πρώτης χρονιάς ισχύω της ε, συνθήκης της Λισαβόνας. Για οργανωτικούς λόγους, αντί να αρχίσει να ισχύει τόσο γρήγορα δεν θα αρχίσει να ισχύει παρά τον επόμενο Απρίλιο. Αλλά εμείς θα πρέπει να κρατήσουμε σαφές ότι θα πρέπει αμέσως να ξεκινήσει η πρωτοβουλία και όχι να ξεκινήσουμε μία νέα διαδικασία σκέψης γύρω από την πρωτοβουλία πολιτών για την ε, μεταρρύθμιση που προτείνουν η κυρία Γκουρμάη και ο κύριος ε, Λαμασούρ ε, εκφράζουν τις ανησυχίες και οι ανησυχίες συγγνώμη, του κυρίου Αλεξάνδερ έχουν νόημα διότι η πρωτοβουλία πολιτών τι προβλέπει ότι μετά από συγκεκριμένη περίοδο λειτουργίας θα πρέπει να προχωρήσουμε στη διαδικασία αναθεώρησης και αυτή η αναθεώρηση θα μας δώσει τη βάση για να προχωρήσουμε σε αλλαγές και αναθεωρήσεις οι οποίες θα είχαν τη θέση τους σε μία έκθεση πρωτοβουλίας. Τώρα, μία έκθεση τρόπολο, ε, ε, πρωτοβουλίας δεν θα είχε κανένα νόημα, διότι μαζί με αυτή τη διαδικασία που έχουμε για να προχωρήσουμε γρήγορα θα δημιουργούσε μόνο σύγχυση. Ο κύριος Μπρόντς. Και μετά κλείνουμε με την απάντηση της κυρίας Γκουρμάη. Ναι. Η πρωτοβουλία πολιτών αναφέρθηκε ως στοιχείο συμμετοχής δημοκρατίας ή τουλάχιστον τρόπο συμμετοχής των πολιτών αλλά στην πραγματικότητα ένας πάρα πολύ ρυθμισμένος και περιορισμένος τρόπος συμμετοχής. Υπάρχουν διάφοροι κανόνες περί του αποδεκτού, δεν πρέπει να είναι για πλάκα μέσα σε εισαγωγικά αυτή η πρωτοβουλία πολιτών. Βέβαια εδώ υπάρχει μια υποκειμενική άποψη, για να το κρίνει κανείς. Δεν πρέπει να είναι κατά των ευρωπαϊκών αρχών, αλλά και εδώ μήπως είναι ένας τρόπος να εμποδίσουμε περαιτέρω αποφάσεις της Ευρωπαϊκή Ένωση Και ο Επίτροπος Σεύκοβιτς έθεσε μια περαιτέρω συνθήκη δεν πρέπει να είναι εναντίον του συμφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ αν είναι υποκειμενικό αυτό. Αυτό θα εμπόδιζε εκπεφρασμένα απόψεις που έχουν να κάνουν με απόψεις οι οποίες είναι κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ακόμα και με αντιπαγκοσμιοποιητικές απόψεις που αντιτίθενται στο φιλελεύθερο πνεύμα που επικρατεί αυτή τη στιγμή. Εγώ θεωρώ ότι μια περιορισμένη δημοκρατία δεν είναι δημοκρατία, είναι απλώς μια κλάκα η οποία έχει ενορχιστρωθεί. Οι πολίτες οι οποίοι δεν συμμετέχουν σε ομάδες πιέσεων ή σε κόμματα σε πολλές χώρες, το να μπορέσουν να συγκεντρώσουν ένα εκατομμύριο υπογραφές αυτό είναι απλοϊκό και υπερβολικά αθώο, πιστεύω. Να νομίζει κανεί ότι μπορεί να γίνει αυτό χωρίς τη συμμετοχή κομμάτων ή άλλων ομάδων πίεση. Κυρία Σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Χαίρομαι που όλοι μελετήσατε αυτές τις δυνατότητες που ανοίγονται με αυτή την πρωτοβουλία πολιτών. Πρέπει να πω ότι υποστηρίζω μια απλή και άμεση προσέγγιση, να μην κάνουμε τα πράγματα πιο δύσκολα για τους πολίτες Νομίζω ότι έχουμε τις τροπολογίες και μπορεί η συνέλευση των Προέδρων των πολιτικών ομάδων να αποφασίσει ποια είναι η καλύτερη δυνατότητα να ακολουθηθεί και αυτό θα δώσει δυνατότητα σε όλους τους συναδέλφους που έχουν διαφορετικές ε, προσεγγίσεις να συμμετάσχουν στην απόφαση για το θέμα αυτό. Εγώ χαίρομαι λοιπόν που υποστηρίζετε αυτή την απλή και διάφανη διαδικασία. Ευχαριστώ. Θέλει κανείς άλλο το λόγο, ναι. Ναι, το θέμα αυτό το είχαμε συζητήσει και με τους υπεύθυνου. είχε συμφωνηθεί ότι τα θέματα τα οποία θα πρέπει να διευκρινιστούν ίσως να είναι λίγο διαφορετικά σε εκτάση, αλλά επί της ουσίας νομίζω είναι πολύ παρόμοια. Είχε συμφωνηθεί λοιπόν ε, να ακολουθηθεί η ίδια μορφή που κρατάμε ως τώρα. Δηλαδή όσοι είχαν εργαστεί ως τώρα για το θέμα αυτό να συνεχίσουν να εργάζονται γι' αυτό και είχαμε πει ότι ενδεχομένως ε, με την Επιτροπή να διαλέξουμε ένα διαφορετικό εργαλείο, είτε δηλαδή ε, αλλαγή του κανονισμού ε, ή έκθεση πρωτοβουλίας. Εγώ θα προτιμούσα έκθεση πρωτοβουλίας, αλλά συμφωνώ και με την άλλη μορφή. Το θέμα όμως είναι να λυθούν και να ε, διευκρινιστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα ανοιχτά θέματα. Αυτά που είπε ο κύριος Σούπλεν για την σύγκρουση των πολιτισμών, αν θέλετε. Νομίζω ότι από διάφορες μελέτες προκύπτει ότι πολλά λειτουργούν όταν υπάρχει καλή ρύθμιση. Αντίθετα, όταν δεν υπάρχει καλή ρύθμιση, συχνά προκαλούνται διαμάχες. Ωραία λοιπόν να γίνει μια περισυλλογή αλλά να ακολουθήσει και μια καλή ρύθμιση μετά. Μου φαίνεται όμως να υπάρχει εδώ ευρύτατη συνένεση. Δηλαδή να ακολουθήσουμε το δρόμο της ε, τροποποίησης του κανονισμού. Και ούτως θα πράξουμε οι εισηγητές στη συνέχεια θα πρέπει να παρουσιάσουν τις τροπολογίες τους και μετά στους συντονιστές θα αποφασίσουμε το πώς θα συνεχίσουμε την πρωτοβουλία. Ωραία. Πάμε στο επόμενο σημείο. Όχι, ναι. Α, ναι, ναι, ναι. το θέμα, η αναθεώρηση. Λάθος, λάθος. Α, πού είναι αλήθεια, πού είναι αλήθεια. Μάλιστα, αυτή είναι η ημερήσια διάταξη. Ακριβώ. Ακριβώς ορίστηκε η εισηγητής για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονία, ο κύριος Νταφ. Πρόκειται για ένα σχέδιο γνωμοδότησης το, για, για την ΑΦΕΤ η οποία θα ψηφίσει στις 12 ε, Νοεμβρίου. Όπως ξέρετε η Κομισιόν έχει ξεκινήσει μια μεγάλη μεταρρύθμιση και γενικά θεωρείται ότι αυτό μπορεί να είναι μια βελτίωση για την πολιτική γειτονία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κύρια έκθεση είναι από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του κυρίου Σιέβετς και του κυρίου Νταβίτ. Υποστηρίζει τη γενική κατεύθυνση της ε, πρότασης της Κομισιόν. Κατά την άποψή μου όμως δεν καταφέρνει να αντιμετωπίσει με τρόπο επαρκή τις θεσμικές απόρριες της ενίσχυσης της ε, πολιτικής γειτονίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτές οι πτυχές είναι τόσο και εσωτερικού χαρακτήρα για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και έχουν και την εξωτερική διμερή και πολυμερή ακόμα πτυχή των σχέσεών μας με τις χώρες αυτές. Χρειάζεται λοιπόν να δημιουργήσουμε ένα πιο σταθερό και ανθεκτικό πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ ημών και των γειτόνων μας. Στο σχέδιο αυτογνωμοδότησης εγώ παρουσιάζω αυτά που θεωρώ ότι πρέπει να είναι τα θέματα τα οποία μας δημιουργούν ακόμα ανησυχίες και προβλήματα. Στην πρώτη παράγραφο αναφέρομαι στον λόγο, στο λόγο ύπαρξης της ε, πολιτικής γειτονίας που είναι να ενισχυθεί η οικονομική και πολιτική ολοκλήρωση μεταξύ ημών και των γειτόνων μας. Η δεύτερη παράγραφος κάνει μια διάκριση των ε, πολυμερών βημάτων όπως είναι η ενωσία τη Μεσόγειο που θα πρέπει κατά την άποψή μου να περιοριστεί σε στρατηγικού χαρακτήρα θέματα και η περιφερειακού χαρακτήρα διμερής και των περιφερειακών διμερών επαφών που είναι σημαντικές για τη βελτίωση της οικονομικής ενσωμάτωσης και της πολιτικής σύνδεσης για τις χώρες οι οποίες εμπλέκονται. για την Ένωση για τη Μεσόγειο θεωρώ μαζί με πολλούς άλλους ότι έχει σχεδιαστεί από άτομα τα οποία δεν είχαν πολύ καλή γνώση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε καταλάβαιναν πολλά και από τη Μεσόγειο. Και ο αντίκτυπός της ε, ήταν μάλλον αντιπαραγωγικός και πρέπει να υπάρξει μία εκβάθρον αναδιάρθρωση και ανασχεδιασμός της Ένωσης και τη Μεσόγειο αν πρόκειται να επιβιώσει εκεί δεν είναι ιδιαίτερα στεναρή η θέση της ε, Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και γι' αυτό νομίζω ότι η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων θα πρέπει να τονίσει την ανάγκη να υπάρχει μια καλύτερη <clears throat> διαχείριση από την ευρωπαϊκή πλευρά της ε, Ένωσης για τη Μεσόγειο να ενταχθεί στα πλαίσια της συνθήκης και να έλθει κάτω από την αιγίδα της υπάτης εκπροσώπου και της υπηρεσίας εξωτερικών σχέσεων. Στην παράγραφο 4 εφιστώ την προσοχή στο αυξανόμενο άχθος για το Κοινοβούλιο του πολυπολαπλασιασμού των διμερών και πολυμερών μορφών συνεργασίας σε κοινοβουλευτικό επίπεδο. Νομίζω ότι με μεγάλη χαλαρότητα αποφασίσαμε να διωγγώνουμε συνέχεια τον αριθμό των διεθνών αυτών κοινοβουλευτικών σωμάτων τα οποία δημιουργούμε, <clears throat> ιδίως στη γειτονιά μας, αλλά όχι μονάχα στη γειτονιά μας και πρέπει να είμαστε λιγάκι πιο επιλεκτικοί όταν συμφωνούμε να έχουμε μελλοντική περαιτέρω ανάπτυξη των διακοινοβουλευτικών αυτών επαφών και βημάτων που στοχεύουν στη συνεργασία. Πέμπτη παράγραφος. Εκεί ζητώ από την Κομισιόν να είναι σαφέστερη σε σχέση με την έννοια του αναβαθμισμένου καθεστώτος που έχει δοθεί στο Μαρόκο τώρα που γίνεται ουσιαστικά ένα κίνημα απελευθέρωσης από τις δεσποτικές κυβερνήσεις στο Μασφέκ και στο Μαγαέπ είναι σημαντικό η ευρωπαϊκή πλευρά να δείξει μεγαλύτερη ευκαινησία και μεγαλύτερη σαφήνεια σε σχέση με το τι μπορεί να προτείνει σε σχέση με τις πολιτικές και θεσμικές μας σχέσεις με τις αραβικές χώρες. Και το να καταφύγουμε, όπως κάναμε στο παρελθόν, σε αμφίσιμες έννοιες, όπως το αναβαθμισμένο καθεστώς, αυτό δεν μας βοηθάει ιδιαίτερα. Έκτος, έχουμε να κατανοήσουμε ότι έχουμε δημιουργήσει δύο εργαλεία τα οποία στοχεύουν να κάνουν ακριβώς το ίδιο. Με διπλή επιβάρυνση στον προϋπολογισμό μας. Και νομίζω ότι η Επιτροπή μας θα πρέπει να επιμείνει να γίνει μια διάκριση και από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων με μια διάκριση μεταξύ, μεταξύ του ρόλου του Ευρωπαϊκού Εργαλείου για τη Δημοκρατία και του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Δημοκρατία, καταπιστεύματος για τη Δημοκρατία. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να έχουμε τόσες επικαλύψεις και συγχύσεις μεταξύ των δύο αυτών οργάνων. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μας εξυπηρετεί. Θα μπορούσε να υπάρχει μια διάκριση μεταξύ των δύο που να είναι σαφής. Μέχρι στιγμής η Κομισιόν και η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων δεν έχουν προσεγγίσει το θέμα της σαφέστερης διάκρισης. Και εν τέλει υπάρχει η πρόταση του ότι θα πρέπει να δείξουμε μεγαλύτερη συνεκτικότητα και συνέπεια σε μακροπρόθεσμο επίπεδο σε σχέση με την σταθεροποίηση του πολιτικού και θεσμικού μας ρόλου με τρίτες χώρες, χώρες που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει μια ρευστή κατάσταση στον περιγυρό μας και λόγω αυτού θα ήταν αμοιβαία εποφελές το να έχουμε μια πιο άμεση κατεύθυνση και για μας και για τους γειτονές μας προς μια μορφή σχέσης εταιρικού χαρακτήρα, σχέση σύνδεση που να είναι αποδεκτή και για μας και για αυτούς. Και είναι εξάλλου πολύ επίκαιρο το γεγονός ότι στην επόμενη μεταρρύθμιση των συνδικών που θα ξεκινήσει το, την επόμενη άνοιξη είναι απαραίτητο να θέσουμε στην ημέρησια διάταξη της συνέλευσης που θα προετοιμάσει τη νέα συνθήκη μία πρόταση να υπάρξει και ένα νέο πλαίσιο για επίσημη σχέση συνδεωμένης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρας, το οποίο θα καλύψει τέσσερα είδη κρατών. Πρώτα, τα κράτη αυτά τα οποία δεν εκπληρούν τα κριτήρια της συνθήκης για να είναι ευρωπαϊκά κράτη, και επομένω δεν μπορούν ποτέ να γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δεύτερη κατηγορία αφορά κράτη τα οποία ενώ θεωρητικά θα μπορούσαν να ζητήσουν να γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφασίζουν ότι δεν θέλουν να κάνουν μια τέτοια αίτηση εισδοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η τρίτη κατηγορία, η κατηγορία για τις χώρες που προσπαθούν, προσπαθούν αλλά δεν τα καταφέρνουν οι χώρες δηλαδή για τις οποίες η εκπλήρωση των κριτηρίων της Κοπενχάγης και όλων των άλλων κριτηρίων αποτελεί μια πολύ μεγάλη πρόκληση που δεν μπορούν προς το παρόν να την αντιμετωπίσουν και που χρειάζονται μια εξασφαλισμένη θέση ώστε για ένα χρονικό διάστημα μέχρι να μπορέσουν να εξασφαλίσουν την εκπλήρωση των ε, κριτηρίων θα χρειαστούν κάποιο χρόνο, μιλάω εδώ πέρα κυρίως για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, αλλά υπάρχει και μια τέταρτη κατηγορία. Και αυτή αφορά ένα κράτος μέλος, το οποίο είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θεωρεί ότι το βήμα που πρέπει να κάνει προς την κατεύθυνση μιας ομοσπονδιακής Ευρώπης είναι κάτι το οποίο είναι υπερβολικό, δεν θέλει να το, να το κάνει και αποφασίζει να αποσυρθεί σε μία μορφή σύνδεσης που δεν του αποστερεί όλα τα λειτουργικά στοιχεία σχέσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να υποστηρίζει το στόχο της ε, οικονομικής ολοκλήρωσης και της πολιτικής εταιρικής σχέσης, αλλά θέτει εαυτόν θα βγει έξω από το ομοσπονδιακό γήπεδο ούτως υπήν. Θεωρώ ότι όλα αυτά βέβαια είναι αρκετά ουσιαστικά σε επίπεδο γνωμοδότησης. Πιο ουσιαστικά από ότι περιμένει κανείς από μια γνωμοδότηση αυτού του είδους. Στα πλαίσια μιας γνωμοδότησης στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Αλλά λόγω της σημασίας του, της έκθεσης της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων για την ε, πολιτική γειτονία και λόγω της αστάθειας και του πυρετόδους και εργόδους χαρακτήρας των καιρών που περνάμε, νομίζω ότι αξίζει το κόπο να να φτάσει σε μια χρονοδότηση. Συγγνώμη που δεν μπόρεσα να ακούσω όλα αυτά που είπε ο συνάδελφος Νταφ. Είχα κάποιες υποχρεώσεις και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Γκέρα εδώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Νταφ για το σχέδιο γνωμοδότησής του που μας έχει παρουσιάσει σε σχέση με την έκθεση πρωτοβουλίας της Επιτροπής Εξωτερικών Θεμάτων. Κατά την άποψή μου, ορισμένα στοιχεία αυτής της γνωμοδότησης είναι άξια υποστήριξης. Υπάρχει ένα σημείο για το οποίο εγώ θα ήθελα να σκεφτούμε λίγο περισσότερο. Και υπάρχει και μια τρίτη πτυχή. Υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία μου δημιουργούν κάποιες αμφιβολίες είτε σε μένα είτε στην πολιτική μου ομάδα, στη σοσιαλιστική ομάδα. Από τα θέματα τα οποία πρέπει να τα εξάρω θετικά και να τα υποστηρίξω περιλαμβάνουν την προσέγγιση υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την υπεράσπιση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στην πολιτική γειτονία μας. Είναι σημαντικά όλα αυτά γιατί πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι στις σχέσεις μας με τους γείτονες δεν έχουμε πάντα δώσει την απαραίτητη έμφαση στα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας. Και επίσης, η όθηση που ζητά ο κύριος Νταφ να δοθεί από το Κοινοβούλιο για να υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή του Κοινοβουλίου στην πολιτική γειτονία είναι και αυτό κάτι το οποίο αξίζει να το υποστηρίξουμε. Αλλά όπως είπα προηγουμένως υπάρχει ένα σημείο το οποίο χρειάζεται περισσότερη σκέψη και αυτό αφορά την Ένωση για την Μεσόγειο. Σύμφωνα με την ισπανική εκδοχή του κειμένου. Εγώ δύο μόνο το ισπανικό κείμενο διάβασα. Εδώ βλέπω να υπάρχει μια απόρριψη του εισηγητή της Ένωσης για τη Μεσόγειο ως πρωτοβουλία, ως θεσμό. Εγώ συμμερίζομαι με τον κύριο Ντάφ και νομίζω ότι δεν είμαι μόνος την ε, εντύπωση ότι η σχέση μας με τους γείτονες της νότιας όχθης της Μεσογείου δεν ήταν δεν έχει σταθεί υποδειγματική από πολλές απόψεις. Ζούμε τώρα αυτή την γενική κινητοποίηση της Αραβικής Άνοιξης. Ούτε η σχέση μας με τις χώρες αυτές ήταν μια ιδιαίτερα αποτελεσματική σχέση και υπήρξαν και πολλά σημεία ασυνέχεια σε αυτή τη σχέση. Θυμάται ο κύριος Δάφο στην αρχή της θεσμοποίησης των σχέσεων μας με την ε, Νότια Μεσόγειο ξεκίνησαν το 1995 με τη λεγόμενη διαδικασία της Βαρκελόνης που ενεκρίθη υπό Ισπανική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 1995. Στη συνέχεια όμως η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και η ταραχώδης σχέση μεταξύ της κυβέρνησης του Ισραήλ και των κυβερνήσεων των αραβικών χωρών της Νότιας Μεσογείου ουσιαστικά έχουν μπλοκάρει τις περισσότερες πρωτοβουλίες και τον πολιτικό διάλογο, την ε, επέκταση και των εμπορικών σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών αυτών. Οπότε, εγώ δέχομαι μεν τη διάγνωση που παρουσιάζει ο κύριος ε, Νταφ, ότι η διαδικασία της Βαρκελόνης καταρχήν και η Ένωση για τη Μεσόγειο σήμερα έχουν προχωρήσει πολύ λιγότερο και έχουν μπει πολύ, πολύ λιγότερο σε βάθος από ό,τι θα έπρεπε να είχαν κάνει. Αλλά νομίζω ότι τώρα ακριβώς έχουμε την ευκαιρία να τους δώσουμε μια νέα προσέγγιση. Τονίζω και πάλι. Στο ισπανικό κείμενο, διαβάζοντας το, μπορεί κανείς να καταλήξει το συμπέρασμα ότι ο κύριος Νταφ αυτό το οποίο επιζητεί είναι να εξαφανιστεί από το χάρτη η Ένωση για τη Μεσόγειο. Ενώ εγώ νομίζω ότι πρέπει αντίθετα να εξασφαλίσουμε την ανασογόνηση αυτής της Ένωσης για τη Μεσόγειο για να ανταποκριθούμε ακριβώς στις προσδοκίες που έχουν αναφύει με τη διαδικασία αλλαγής στη νότια οχτή της Μεσογείου. Αυτό λοιπόν είναι ένα σημείο το οποίο θα πρέπει να μας προβληματίσει λίγο περισσότερο και να έχουμε μια διαφορετική διατύπωση στην αρμόδια παράγραφο. Τώρα για το τελευταίο σημείο. Ούτε υποστηρίζω, ούτε στρέφομαι εναντίον αυτού που ανέφερε ο κύριος Σταφ για την επιζήτηση κάποιας φόρμουλας, μιας μορφής σχέσεως σύνδεσης για χώρες οι οποίες ενώ εκπληρούν τις προϋποθέσεις για να είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προτιμούν να μείνουν απ' έξω, προτιμούν μια άλλη μορφή σχέση. Νομίζω όμως ότι πρέπει αυτό να το εξετάσει η ομάδα μου, η σοσιαλιστική ομάδα και θα μπορέσουμε στη συνέχεια σε συζήτηση με τον κύριο Νταφ και μέσω τροπολογιών να παρουσιάσουμε τη δική μας άποψη η οποία να είναι λίγο πιο επεξεργασμένη για το σημείο αυτό. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ κύριο Σέπλιν. Ευχαριστώ πρόεδρε και πάλι. Θα ήθελα να σας ε, μεταδώσω την θέση του ΕΛΚ. Να ξεκινήσω από αυτά που είπε ο Άντριου Νταφ. Ναι, όντω είναι πραγματικά πυρετόδης η εποχή αυτή. Και νομίζω ότι αυτό συνεπάγεται ότι με τους όρους αυτούς είναι δύσκολο να κάνουμε τέτοιες προβλέψεις, γιατί αν αποκατεβαίνει η θερμοκρασία είτε με βαθμούς Φαρενάιτ, είτε με βαθμούς Κελσίου, θα, θυμάτε, θα θυμάστε ότι παλιά θα χρησιμοποιήσετε κι εσείς. Υπό τους όρους λοιπόν αυτούς είναι δύσκολο να ε, δημιουργήσουμε ένα σταθερό πλαίσιο, όπως ανέφερε ο κύριος Νταφ. Άρα αυτό σημείο εκκίνησης θα πρέπει να το πάρουμε και άρα θα πρέπει να κοιτάξουμε πού μπορούμε να βρούμε πιο ισχυρές ε, ρυθμίσεις, θεσμικές ρυθμίσεις. Υπάρχει κάποιο θεσμικό έλλειμμα άλλωστε στην περιοχή αυτή και να αναφερθώ εδώ πέρα στην ε, υπηρεσία για την κοινωνία των πολιτών που βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης και τέτοιου είδους ρυθμίσεις. Δεν είμαι βέβαιος τώρα το τι σημαίνει η εναρμόνιση αξιών σε επίπεδο ΟΗΕ. Τι σημαίνει αυτό. Δεν είμαι βέβαιος ότι αποδεχόμαστε όλες τις αξίες του ΟΗΕ. Νομίζω ότι υπάρχει διαφορά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ΟΗΕ ίσως θα έπρεπε να εναρμονίσει τις δικές του αξίες με τις δικές μας, αλλά αυτό αποτελεί διαφορετικό ζήτημα. Στο δεύτερο σημείο τώρα λέμε νομίζω ότι θα πρέπει να φερθεί πιο έντονα η ανατολική διάσταση. Αυτό θα πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα σε σχέση με τη σημερινή κατάσταση. Στο σημείο 3 θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ έντονη η διατύπωση. Ανεπαρκή σύλληψη, κακή εκτέλεση, ενδεχομένως αντιπαραγωγική. Αυτό πραγματικά μας δυσκολεύει. Δεν ξέρω αν θα τα αποδεχτούμε για το επόμενο σημείο τώρα. Για την ε, Euronest και την Ευρωμεσογειακή Κοινοβουλευτική Συνέλευση. Ξέρουμε ότι η Euronest δεν ε, λειτουργεί τέλεια, αλλά αξίζει τον κόπο. Έχει συνέλθει δύο φορές νομίζω ως τώρα με σημαντικές δυσκολίες, αλλά θεωρώ παρά τις δυσκολίες αυτές ότι θα πρέπει να εμείνουμε. Στο τελευταίο τώρα σημείο, κοιτώντας την ιδέα της νέας ε, κατηγορίας χωρών με τις οποίες υπάρχει συνεργασία, θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ το θέμα της παρουσίασης, του image αν θέλετε. Νομίζω ότι σε κάποιες χώρες αυτό θα φανεί ότι είναι δευτεροκλασσάτες. Να δημιουργηθεί λοιπόν θεωρώ ένας ευρωπαϊκός πολιτικός χώρος. Αυτό θα ήταν πλέον κατάλληλο. Κάπως έτσι να το ονομάσουμε και θα πρέπει να διασφαλίσουμε και αυτό είναι ουσιώδες ότι θα συμμετάσχουν η Ελβετία και η Νορβηγία γιατί αυτό θα δώσει κύρος στα μάτια χωρών τις οποίες αναμφίβολα έχετε υπόψη σας. Και νομίζω ότι θα πρέπει να είναι επίσης σαφές, όσο πιο σαφές γίνεται, ότι αυτό το καθεστώς δεν σημαίνει ότι παγιδεύεται κάποια χώρα μονίμως σε αυτό το χώρο. Όχι, θα υπάρχει δυνατότητα προώθησης. Αυτό θα πρέπει να είναι σαφές. Μου αρέσει η ιδέα τροχιάς, αν θέλετε, στάθμευσης για κάποιες χώρες. Κάποιες από τον οποίων θα είναι ίσως, ε, θα έχουν λάβει ένα όχι ως απάντηση. Εκεί θα ήταν άλλωστε και το Ηνωμένο Βασίλειο στη δεκαετία του 60. Πριν το 73. Άρα δεν είμαστε κάθετα εναντίον αυτής της ρύθμισης, αλλά θα πρέπει να διατυπωθεί με τέτοιο τρόπο που να προωθεί και όχι να καθυστερεί την εφαρμογή των στόχων μας. Thank you, um, Σε ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Ντάφ στο θέμα για το... την γνωμοδότηση αυτή. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Κάνα δύο ερωτήσει, επιτρέψτε μου. Σε ό,τι αφορά την Ένωση για τη Μεσόγειο, αναφέρεται ότι η, η αρμοδιότητα είναι της ύπατη εκπροσώπου. Αυτό φαντάζομαι είναι λογικό. Αλλά εμεί ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε ασφαλώ μια διαρκή συζήτηση με του εκπροσώπους μα. Αυτό δεν ισχύει με τα εθνικά κοινοβούλια τα οποία εκπροσωπούνται στην Ένωση για τη Μεσόγειο. Κοιτώντα λοιπόν αυτή την αρμοδιότητα, αν τη δώσουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αποκλειστούν τα εθνικά κοινοβούλια από τη συζήτηση, ενώ εμείς θα έχουμε αυτή την δίωδο επικοινωνίας με την Αντιπρόεδρο. Άρα υπάρχει θεωρώ ένα πρόβλημα. Θα πρέπει να κοιτάξουμε πώς θα διατηρηθεί η εμπλοκή των Εθνικών Κοινοβουλίων σε ό,τι αφορά τη συζήτηση για την Ένωση για τη Μεσόγειο και κατά δεύτερον φυσικά με ενδιαφέρει ιδιαίτερα το θέμα της ε, ένταξης αυτής. Ε. Τρεις κατηγορίες, τέσσερις κατηγορίες ανέφερε ο κύριος Νταφ σε ό,τι αφορά το καθεστώς των ε, τρίτων χωρών. Θα μπορούσαμε να ορίσουμε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια ποια θα είναι ο στόχος αυτός, αυτής της ένταξης, αυτής της συμμετοχής. Και θα υπάρχουν μεμονωμένες διαπραγματεύσεις αναχώρα. Ή κάθε κατηγορία θα περιλαμβάνει ένα ταυτόσιμο πακέτο για όλες τις χώρες. Για διασφαλώς υπάρχουν και διαφορετικοί όροι για κάθε, χώρες, για κάθε χώρα. Αυτές λοιπόν οι ερωτήσεις μου πληροφοριακές και θα πρέπει να τι διευκρινίσουμε. Ιδιαίτερα με απασχολεί αυτό με τα εθνικά κοινοβούλια, να μην αισθανθούν ότι τα κλειδώνουμε απ' έξω, γιατί δεν θα δεχτούν ποτέ, φαντάζομαι, να κλείσει το φόρουμ αυτό, αν δεν λάβουν κάποιον άλλο τρόπο άσκηση επιρροή. Ευχαριστώ κύριε Μέσερ Σμιτ. Ο κύριος Ένιου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μου είπαν ότι έχω το δικαίωμα να λάβω το λόγο και νομίζω ότι αυτά που είπε ο κύριος Δάφ είναι πολύ ενδιαφέροντα. Γιατί <clears throat> είπε ότι θεωρεί ότι την Άνοιξη θα υπάρξει η ευκαιρία να τροποποιηθούν οι συνθήκες της Λισαβόνης. Αυτό φαίνεται να αντιβαίνει αυτά που είπε στην, ε, στη, στο κομματικό συνέδριο των συντηρητικών ο πρόεδρος της Μεγάλης Βρετανίας που είπε ότι δεν υπάρχουν, δεν υπάρχουν προοπτικές τροποποίησης των ε, συνθήκων μια συνδεόμενη σχέση μέλους είναι πολύ ενδιαφέρουσα και είναι η τέταρτη κατηγορία που ανέφερε ο κύριος Τάφ. Τα κράτη-μέλη που θεωρούν ότι του ζορίζει υπερβολικά η συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρω σε ποιον αναφέρεται, <clears throat> ίσως αναφέρεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, που αυτό το θέμα της συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα καυτό θέμα τώρα. Ναι, ας πούμε ότι μπαίνουμε σε αυτό το νέο σχήμα ως Ηνωμένο Βασίλειο τίθενται δύο ερωτήματα. Αυτή η κατηγορία θα συμμετέχει οικονομικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντισταθμίσει το προνόμιο του να είναι συνδεόμενο μέρος. Και δεύτερον, θα εφαρμόζονται οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτούς ιδίως στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής και της μετανάστευσης. Ευχαριστώ. Ο συνάδελφος Δάπια να απαντήσει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς που έχουν κάνει παρατηρήσεις για την ε, παρουσίαση αυτή. Οι κανόνες για τη γνωμοδότηση περιορίζουν τον, ε, το μήκος της ε, γνωμοδότησης και δεν επιτρέπουν αιτιολογική έκθεση για τη γνωμοδότηση. Αλλά για να εξηγήσω καλύτερα τη στάση μου για την Ένωση της, για τη Μεσόγειο, θα ήθελα να στείλω μια έγγραφη, ένα έγγραφο υπόμνημα στον πρόεδρο της Επιτροπής μας και να το διαβιβάσει σε όλους τους ε, ενδιαφερόμενους για να δει γιατί υπάρχει αυτή η επικριτική μου στάση σε σχέση με όλα αυτά που έχουν λάβει η χώρα μέχρι τώρα. Δέχομαι ότι ο κύριος Γκερέρο έθεσε το ερώτημα του αν θέλω να διαγραφεί τελικά από το χάρτη η Ένωση για τη Μεσόγειο. Όχι, δεν είναι αυτός ο στόχος μου. Αλλά για να επιβιώσει πράγματι πρέπει να μεταμορφωθεί και θα ήθελα να μεταμορφωθεί αυτή η Ένωση για τη Μεσόγειο. Υπάρχει ένα δυναμικό το οποίο δεν έχει εκπληρωθεί μέχρι στιγμής. Αλλά για να μπορέσει να γίνει πραγματικότητα αυτό το δυναμικό θα πρέπει να τεθεί μέσα σε κάποια πειθαρχία. Την πειθαρχία της κοινή εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, κάτι το οποίο δεν ισχύει αυτή τη στιγμή. Αλλά μπορώ σε ένα έγγραφο σημείωμα να τα εξηγήσω αυτά πολύ καλύτερα. Για τον κύριο Σέφριν. η ευθυγράμμιση των αξιών για την οποία αναφέρθηκα είναι ευθυγράμμιση αξιών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των γειτόνων της. Μέσα στο Ηνωμένο, στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Αυτό ίσως είναι κάπως ε, προχωρημένο για ορισμένους. Δεν ε, μπορεί κανείς να έχει μία ταυτότητα απόψεων σε, όλες τις, ε, σε όλους τους φορείς και τα βήματα του ΟΗΕ, αλλά το να υπάρχει μια κοινή αντιμετώπιση για τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, για το κράτος δικαίου, για τον αγώνα κατά της διαφθοράς, όλα αυτά το να γίνονται με κοινή συμφωνία μεταξύ ημών και των γειτόνων μας στα διεθνή φόρα, αυτό μου φαίνεται ότι είναι μια σαφής ε, ιδέα και ένα συγκεκριμένο στόχος προς τον οποίο θα πρέπει να κινηθούμε <clears throat> και να ζητήσουμε από τους συναδέλφους μας στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων να θέσουν στο κέντρο της προσέγγισής τους για τη μεταρρύθμιση της πολιτικής γειτονία. Σε αυτά που είπε ο Μόρτεν Μέσσερ Σμιτ το να υπάρξει μια μνήα στη λειτουργία των Εθνικών Κοινοβουλίων στην Ένωση για τη Μεσόγειο. Ναι, θα το περιλάβω και αυτό στην επιστολή μου προς τον κύριο Κασίνη. Αλλά αυτή τη στιγμή τα Εθνικά Κοινοβούλια είναι τόσο απόκληρα αυτή τη διαδικασία όσο είμαστε κι εμείς. Δηλαδή η κοινοβουλευτική διάσταση του κοινοβουλευτικού ελέγχου της Ένωσης για τη Μεσόγειο είναι πάρα πολύ περιορισμένη αν είναι ορατή καν, αν υπάρχει καν. Και συμφωνώ με αυτά που λέτε πρέπει να βελτιωθεί. Για την παράγραφο 7. Ναι, πολλά ερωτήματα πρέπει να τεθούν και να απαντηθούν. Δεν έχω εδώ τις απαντήσεις. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο θέλω τα σχόλιά σας γιατί αυτή τη στιγμή μόνο μέσα στο πλαίσιο που αφορά την Κομισιόν, τους Πρωθυπουργού, τα Εθνικά Κοινοβούλια και μέσα σε αυτούς τους Πρωθυπουργού είναι και ο ίδιος ο κύριος ο Κάμερον αλλά που περιλαμβάνει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μόνο μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο μπορούμε να αποφασίσουμε και να σχηματοποιήσουμε το τι θα σήμαινε μια τέτοια σχέση σύνδεσης. Και κύριε Σέπλιν, μπορώ να φανταστώ μια τέτοια σχέση να περιλαμβάνει την Νορβηγία και την Ελβετία. Δεν θα είναι αυτό το οποίο λέγαμε παλιά μια προνομιακή εταιρική σχέση. Μια ορολογία που εμένα ποτέ δεν μου άρεσε μου φάνηκε ότι ήταν κάπως πατερναλιστικού χαρακτήρα. Δεν πρέπει να υπάρχει μια πατερναλιστική απόχρωση σε μια τέτοια σχέση. Θα πρέπει να είναι λειτουργική και θα πρέπει να είναι στεγανή σε νομικούς όρους με σαφείς οικονομικούς στόχους και πολιτικούς στόχους. Αλλά όχι τους στόχους κατά ανάγκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωραία όλο τη συζήτηση για την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας. Εγώ προτείνω να ψηφίσουμε 24 Δεκάτου, εάν συμφωνείτε, 24 Οκτωβρίου. Αυτό σημαίνει ότι έχετε προθεσμία για τις τροπολογίες 11 Οκτωβρίου στις 9 το πρωί. Σύμφωνοι. Πάμε στο επόμενο σημείο που είναι η τροποποίηση της πράξης περί της εκλογής των εμμελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρόκειται για ακαμφόδες θέμα, το συζητήσαμε και το θέμα αναβλήθηκε κατά την προηγούμενη ολομέλεια του Ιουλίου και θα μας παρουσιάσει τώρα ένα δεύτερο σχέδιο ο κύριος Νταφ δεύτερο σχέδιο για την εκλογική μεταρρύθμιση. Μάλιστα. Επαναρχόμαστε λοιπόν στο θέμα αυτό. Η συζήτηση στην Ολομέλη τον Ιούλιο ήταν και εκτενής και ε, έντονη. Και μετά ακολούθησε και συζήτηση. Μάλλον είχε προηγηθεί η συζήτηση στην ΑΦΚΟ. Υποσχέθηκα ότι θα λάμβανα υπόψη την κριτική, την επικοτομητική κριτική που ασκήθηκε στην πρώτη έκθεση της Επιτροπής. Άρα έχετε πλέον ενώπιόν σας μια δεύτερη έκθεση. Να περιγράψω τις βασικές αλλαγές, αν θέλετε. Νομίζω από πλευράς χαρακτήρα το έγγραφο πλέον μοιάζει πιο πολύ με έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας. οι προτινόμενες τροπολογίες που ήταν αρχικά στο παράρτημα 3 πλέον δεν συμπεριλαμβάνονται. Βρίσκονται φυσικά στο αρχείο, αλλά δεν συμπεριλαμβάνονται στο τρέχον πακέτο. Νομίζω ότι αυτό θα απλοποιήσει τα πράγματα. και νομίζω ότι σε όσους είναι καινούργοι στο θέμα αυτό θα δώσει ε, ένα λόγο να είναι πιο ήρεμη. Προτείνω να ενισχυθεί και κλείνει το μικρόφωνο του μιλητή. Προτείνω λοιπόν να ενισχυθεί ο ρόλος και η εντολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά τον διάλογο με το Συμβούλιο. Βλέπετε λοιπόν στην παράγραφο 11 τη σχετική πρόταση του ψηφίσματος. αφαίρεσα από την πρώτη παράγραφο την αναφορά στο χρονοδιάγραμμα. Επειδή εκφράστηκε ένα επιχείρημα με το οποίο δεν συμφωνούσαμε, αλλά το άκουσα πάρα πολύ έντονα στην Ολομέλεια, ότι το χρονοδιάγραμμα για τη μεταρρύθμιση της διαδικασίας ήταν λανθασμένο η χρονική συγκυρία. Για τους λόγους που σας είχα εξηγήσει, ο ορισμός της οικονομικής διακυβέρνησης θα έλεγα ότι επιτείνει το εγχείρημα, το επιχείρημα για την μεταρρύθμιση της εκλογικής διαδικασίας για το Κοινοβούλιο. Για την ενίσχυση δηλαδή της πολιτικής νομιμότητας του Κοινοβουλίου. Αλλά όπως και να έχει, προκειμένου να μην προκαλέσω πανικό, αφαίρεσε, εν πάση περιπτώσει, τη συγκεκριμένη αναφορά στο 2014. Αυτό ασφαλώς δεν σημαίνει ότι θεωρώ ότι θα πρέπει να μείνουμε άπραγοι μέχρι τότε, μέχρι το 2014. Ασφαλώς και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να ασκήσουμε πιέσεις. Με κατηγόρησαν ότι δεν κατάφερα να κάνω μελέτη οικονομικού αντικτύπου σε ό,τι αφορά τις προτάσεις. Συμπεριλαμβάνω λοιπόν πλέον και μία πρόταση, μία αναφορά στο κόστος. προκειμένου να παραμείνει στα σημερινά πλαίσια ο προϋπολογισμός του Κοινοβουλίου. Το κατά πόσον πρόκειται για ανοιχτή ψηφοφορία συγγνώμη, για κλειστό σύστημα ψηφοφορίας ή, μη κλειστό σύστημα ψηφοφορίας συμπεριλήφθηκε ως θέμα προσυζήτηση με το Συμβούλιο. Γιατί είναι διχασμένες οι, απόψει, οι απόψεις στο Κοινοβούλιο. 50-50. Και θα πρέπει λοιπόν να μας βοηθήσουν οι φίλοι μας από το Συμβούλιο. Επίσης, κατά πόσον θα είναι οι 25 βουλευτές να προσθεθούν στο σημερινό αριθμό ή κατά πόσον θα πρέπει να συμπεριληφθούν και αυτό θα πρέπει να συζητηθεί στην Ολομέλεια. συζητήθηκε μάλλον στην Ολομέλεια και το συμπεριέλαβα και αυτό στα θέματα που θα συζητηθούν με το Συμβούλιο. Η έντονη εκτίμηση ότι θα χρειαστεί ένα ε, ευρωπαϊκό κατάλογος εκλογιών για την κοινή Ευρωπαϊκή Έντρα. Το συμπερέλαβα και αυτό ε, ως συγκεκριμένη ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αποφασίσουμε για την ε, προσέγγιση μας. προκειμένου να δοθεί σχετική εντολή. Συζήτησα ιδιαίτερα για την Κροατία, επειδή μετά την πρώτη έκθεση της Επιτροπής συμφωνήθηκε ότι η Κροατία θα προσχωρήσει στην Ένωση και ως εκ τούτου δεν μπορούμε επίσημα να ζητήσουμε επανακατανομή των εδρών. 751 οι έδρες. Θα πρέπει όμως η πρόταση να γίνει από το πλαίσιο αυτό. Και φυσικά διατήρησα αυτή τη φιλοδοξία, αυτή την επιθυμία και την πεποίθηση ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε συμφωνία μετά από τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο επί ενός μαθηματικού τύπου για την διαρκή κατανομή των εδρών στο Κοινοβούλιο. Αυτές λοιπόν είναι οι βασικές αλλαγές που έκανα. Στη δεύτερη αυτή εκδοχή του κειμένου. Τι προτείνω. Το συντομότερο δυνατόν να προχωρήσουμε σε τροποποίηση και έγκριση του κειμένου στην Επιτροπή και αντί να πάμε κατευθείαν στην Ολομέλεια όπως συνέβη την προηγούμενη φορά, να ζητήσουμε από τη διάσκεψη των Προέδρων αυτή τη φορά να κάνει μία ανεπίσημη συζήτηση με την Πολωνική Προεδρία και το Συμβούλιο για να βολιδοσκοπήσουμε ενδεχόμενα προβλήματα και τη δική τους ε, αντίληψη για το τι θα πρέπει να συμβεί στο μέλλον. Θα πρέπει με το Συμβούλιο νομίζω να θέσουμε προτεραιότητες για τα μελλοντικά μας βήματα και αν δεν κάνω λάθος και την άνοιξη βρεθούμε σε φάση πλήρους αναθεώρησης της ε, συνθήκης Φυσικά, οι προτάσεις μας σε ό,τι αφορά την εκλογική μεταρρύθμιση θα βρουν τη θέση τους. parola Fox. After the Fox. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω πρώτο. Συγγνώμη στον κύριο Νταφ, γιατί πρέπει να είμαι κάπου αλλού στις 12 ε, και τέταρτο σε 5 λεπτά δηλαδή. Υπάρχουν θετικά στοιχεία σε αυτή την έκθεση και υπάρχουν και σημεία στα οποία εγώ διαφωνώ μαζί του. Προσωπικά λυπάμαι που χρειάστηκε κάπως να αποδυναμωθεί λιγάκι η φόρμουλα η οποία ήταν ένα από τα σημαντικά στοιχεία της προηγούμενης έκθεσης. Χαίρομαι επίση και για τη συμπέληψη παραγράφου 3 που αφορά το κόστο αυτή τη μεταρρύθμιση και νομίζω ότι οποιασδήποτε αλλαγέ κάνουμε πρέπει να είναι ουδέτερε σε σχέση με το κόστο. Δεν πρέπει να επιβαρύνουμε ακόμα περισσότερο τον φορολογούμενο με κόστο διακυβέρνηση. Και επίση νομίζω ότι η ανάγκη για ένα ευρωπαϊκό ψηφοδέλτιο ε, που εγώ θεωρούσα ότι ήταν τελείω περιττό, ότι είχε αποσύρθει από την έκθεση. Για μένα το βασικό πρόβλημα ήταν και εξακολουθεί να είναι η ύπαρξη 25 βουλευτών που να εκλέγονται σε μια ενιαία εκλογική περιφέρεια. Έχω αντιρρήσει αρχή για το θέμα αυτό. Νομίζω ότι η δυσκολία που αντιμετωπίζετε κύριε Ντάφνη είναι εξή. Προηγουμένω προτείνατε να είναι πρόσθετοι 25 βουλευτέ που θα εκλέγονται σε ευρωπαϊκό ψηφοδέλτιο. Τώρα αφήνει το θέμα αυτό ανοιχτό. Θα δείτε όμω ότι τώρα μια διαφορετική ομάδα βουλευτών θα είναι εναντίον αυτή τη ρύθμιση γιατί αν αφαιρέσετε 25 βουλευτές από το σύνολο και αφαιρέσετε τους βουλευτές που θα πρέπει να πάνε στην Κροατία, ορισμένα μικρά κράτη που θα θυγούν λόγω της φόρμουλάς σας θα είναι εναντίον του να υπάρχουν αυτοί οι πρόσθετοι 25 βουλευτές. Είπατε κύριε Ντάφο θα αντιμετωπίσετε τις κυρίες επικρίσεις προς την εκθεσή σας. Μία επίκριση που δεν αντιμετωπίσατε και αυτό λόγω της δικής σας προσωπικής επιμονής στην παράγραφο 2 και τους πανευρωπαϊκούς αυτούς βουλευτές. Αν θέλετε να περάσει αυτή η έκθεση θα πρέπει να ξεφορτωθείτε την παράγραφο 2. Και νομίζω ότι λόγω αυτής της παραγράφου η έκθεσή σας δεν θα γίνει δεκτή. Φιλικά σας λέω λοιπόν, σβήστε παρακαλώ την παράγραφο 2 αν θέλετε να έχετε μια ελπίδα να περάσει η έκθεσή σας. Και επίσης ανησυχώ λιγάκι για την ε, πρότασή σας να παρακάμψουμε τη συζήτηση στην Ολομέλεια και να περάσουμε κατευθείαν σε μια άτυπη συζήτηση με το Συμβούλιο. Ξέρετε ότι δεν είναι δημοφιλή η παράγραφος 2 και γι' αυτό ίσω δεν θέλετε να υπάρξει ψηφοφορία. Πολύ πιο χρήσιμο θα ήταν να έρθει η έκθεση στην Ολομέλεια, να επιτρέψετε να υπάρξει μια ψηφοφορία για τους 25 υπερεθνικούς υποψήφιους. Και φοβάμαι ότι έχω δίκιο όταν σας λέω ότι δεν θα γίνει δεκτή αυτή η παράγραφος στην Ολομέλεια Ίσως γι' αυτό δεν θέλετε να γίνει ψηφοφορία, αλλά εγώ νομίζω ότι πρέπει να γίνει μια συζήτηση για το αν θέλουμε να έχουμε τους πανευρωπαϊκούς αυτούς βουλευτές. Δεν νομίζω ότι είναι χρήσιμη, δεν νομίζω ότι η Ολομέλεια θα τους δεχτεί. Η τελευταία φορά που συζητήσαμε την έκθεση DAF δεν έγινε ψηφοφορία. Έγινε ψηφοφορία γιατί η συνέλευση των Προέδρων δεν μπορούσε να αντέξει την ιδέα μιας, ε, μιας πρότασης η οποία θα υποστήριζε μεγαλύτερη ευρωπαϊκή υπο, ε, ολοκλήρωση, αλλά δεν θα το δεχόταν η Ολομέλεια. Εγώ νομίζω ότι είναι θέμα σεβασμού της δημοκρατίας. Δεν μ' αρέσουν οι άτυπες συζητήσεις με το Συμβούλιο. Είναι καλύτερη η έκθεση αυτή από ό,τι ήταν στο παρελθόν, αλλά έχω ακόμα αντίρρηση για την παράγραφο 2 και εγώ θα ζητήσω να υπάρξει συζήτηση στην Ολομέλεια για να μπορέσουν οι βουλευτέ να εκφράσουν τι απόψει του για αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Ευχαριστώ. Ο Σέπλινγκ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε και να ευχαριστήσω και πάλι τον κύριο Ντάφ. Νομίζω ότι συμφωνώ μαζί του όταν λέει ότι πάμε πάλι από την αρχή. Το έχουμε συζητήσει άλλωστε πολύ εκτενώς το θέμα εδώ στην Επιτροπή και σε άλλα φόρα. Πολλά έχουν συμπεριληφθεί στην έκθεση την αναθεωρημένη με τα οποία συμφωνεί το ΕΛΚ, αλλά για να επανέλθουμε και στην προηγούμενη συζήτηση που είχαμε σήμερα το πρωί πυρετώτες η εποχή που διανύουμε και αυτό δημιουργεί προβλήματα. Ερωτώ λοιπόν και όχι μόνο ρητορικό πώς μπορεί αυτή η μεταρρύθμιση να λάβει την υποστήριξη των πολιτών της Ευρώπης στην παρούσα φάση ή εν πάση περιπτώσει μια πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο. Αμφιβάλλω, όπως είδαμε το καλοκαίρι, δεν είμαι βέβαιος ότι έχουν αλλάξει και τόσα. Κατά πόσον θα γίνει πλήρης αναθεώρηση την άνοιξη της συνθήκης, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά στην παρούσα φάση δεν βλέπω να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Και επίσης ε, πρέπει να σας πω ότι θεωρώ ότι η διαδικασία αυτή είναι μάλλον πιο μακροπρόθεσμη από ό,τι προκύπτει από την έκθεση και νομίζω ότι αποτελεί ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση μεν, το γεγονός ότι δεν συμπεριλαμβάνεται το 2014 ως ημερομηνία αναφοράς, γιατί πρόκειται για πολύ πιο μακροπρόθεσμη διαδικασία. Το ΕΛΚ υποστηρίζει την όλη ιδέα, αλλά και πολλά μπορούμε να κάνουμε για να υποστηρίξουμε τις αλλαγές που προτείνονται περί πανευρωπαϊκού ψηφοδελτίου. Αλλά αυτό θα σήμαινε, θεωρώ, μία περίοδο περισυλλογής, μία ανανέωση της όλης συζήτησης, όπως ε, κατά την πάροδο του χρόνου και όπως θα αλλάξουν και οι πυρετόδους εποχής που ζούμε. Και αυτό σημαίνει, φαντάζομαι, ότι θα πρέπει εκ νέου να θερμομετρήσουμε την κατάσταση σε κάποιο χρονικό διάστημα για να δούμε μήπως τότε θα υπάρξει υποστήριξη. Νομίζω ότι αυτός ο πραγματισμός ε, είναι που χρειάζεται και ίσως να αντίκειται αυτό στις αρχές. Αλλά η άποψή μου και η άποψή του ΕΛΚ είναι ότι θα είναι κρίμα να χάσουμε το σύνολο του κειμένου αν βιαστούμε, αν θέλετε, υπερβολικά. Άρα, τι να σας πω, προτείνω να είμαστε σόφρονες. Eh, Ο κύριος Χέφνερ. Πιστεύω ότι ορισμένες φορές πρέπει να προχωρήσουμε πράγματι προς τα εμπρός. Θα πρέπει να έχουμε το θάρρος τουλάχιστον για να το κάνουμε αυτό, να κάνουμε σημαντικά βήματα προς τα εμπρός και να αναπτύξουμε περισσότερο την Ευρώπη. Δεν νομίζω ότι θα καταφέρουμε να έχουμε μεγάλη υποστήριξη από τους πολίτες μας όταν απλώς προχωρούμε με βήμα σημειωτό. Ο κύριος ε, Νταφ δεν είναι νέο μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχει μακρά ιστορία, έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα για να μπορέσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να πάρει πιο ευρωπαϊκό χαρακτήρα και είναι καλή πρότασή του αυτή για Ευρωπαίους υποψήφιους που εκλέγονται σε ένα ευρωπαϊκό ψηφοδέλτιο. Αυτό είναι σημαντικό να μην υπάρχουν μοναχα βουλευτές οι οποίοι εκπροσωπούν μονάχα τα κράτη-μέλη τους. Είναι καλό να είναι πολίτες ενός κράτους μέλους οι οποίοι εκλέγονται ως Ευρωπαίοι βουλευτές. Αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο της πρότασής του. Έχει λοιπόν, χωρίς να ακυρώσει τα άλλα στοιχεία της συμμετοχής των Ευρωβουλευτών, είναι ένα στοιχείο που κάνει πιο ευρωπαϊκές τις ευρωπαϊκές εκλογές. Αναγκάζει και τα κόμματα να έχουν και κάποιο ευρωπαϊκό χαρακτήρα στην προεκλογική του εκστρατεία. Τα κόμματα λοιπόν περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν θα κάνουν ευρωπαϊκού χαρακτήρα συζητήσεις, θα μπορούν να συζητήσουν περισσότερο για αυτές τις λίστες και αυτό για μένα είναι ένα πολύ καλό και λογικό βήμα. Θα ήταν ίσως καλύτερα τουλάχιστον από την άποψη της δικής μου ομάδας να μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Ίσως η δική μου πολιτική ομάδα ήταν αυτή που υποστήριξε περισσότερο αυτή την έκθεση, ακόμα περισσότερο από ό,τι και οι φιλελεύθεροι στους οποίους ανήκει ο Άντζου Ντάφ, γιατί θεωρούμε ότι αυτό είναι μια καλή κίνηση προς την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας και της Δημοκρατικής Ευρώπης. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι <clears throat> βελτίωση αυτό το νέο κείμενο, όχι γιατί εγώ συμφωνώ με όλα αυτά τα οποία αναφέρονται στο κείμενο, αλλά γιατί θεωρώ ότι η πρόταση αυτή του Άντρου Νταφ θα ξεπεράσει πολλές αντιδράσεις μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όταν δουν ότι το κείμενο έχει αντιμετωπίσει πολλές από τις αντιρρήσεις που είχαν διατυπώσει στο παρελθόν. Αυτό το οποίο προτείνει τώρα ο Άντρου Ντάφ είναι να ξεκινήσουμε μια σύνολη διαδικασία με, ανοιχτό, με ανοιχτή έκβαση αλλά και με μια σαφή στοχοθεσία για να μπορέσει να υπάρξει κάποτε αυτή η ευρωπαϊκή λίστα και επίσης αναφέρει ορισμένες πολλές λογικές ε, προτάσεις για την εκλογή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως παραγωγικά το να γίνεται νωρίτερα, να γίνεται το Μάιο και όχι τον Ιούνιο. Έχει μια σαφή λοιπόν υποστήριξη από μένα. Ο συνάδελφος Φόξ δεν είναι πια παρόν, αλλά είχε πει προηγουμένως ότι το θέμα αυτό για τους 25 αν θα είναι απ' έξω από τους 751 ή μέσα στους 751, στην πρώτη περίπτωση θα αύξανε τον αριθμό των βουλευτών, θα υπάρξει μια αντίσταση λοιπόν από πολλούς, αλλά είπε ο Ασλουφόξ ότι αν είναι μέσα στους 751, δεν θα υπάρξει αντίρρηση για λόγους πρόσθετου κόστους, αλλά θα υπάρξει αντίδραση από αυτούς που θα φοβηθούν ότι αυτό θα μειώσει την εκπροσώπηση των μικρότερων και μεσαίων κρατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ μπορώ να σας πω ότι υπάρχει μια πολύ απλή λύση για να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα και να ξεπεραστεί αυτή η αντίρρηση. Αυτή είναι η πρόταση την οποία έχω υποβάλει στο παρελθόν. Δηλαδή, να υπάρξει ένας απλός κανόνας ότι δηλαδή αυτοί οι βουλευτές που εκλήγονται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο θα υπολογιστούν και στον αριθμό εντολών που αντιστοιχούν σε κάθε κράτος. Δηλαδή δεν θα αλλάξει καθόλου η εθνική σύνθεση των ε, ευρωβουλευτών λόγω της πρόθεσης αυτής. Αυτό είναι ένα σύστημα το οποίο ισχύει σε ορισμένα ε, εθνικά εκλογικά συστήματα Υπάρχει το σύστημα αυτό στη Γερμανία, πραγματικά την Ομοσπονδιακή Γερμανία, όπου ο πολίτης έχει δύο ψήφους. Η πρώτη ψήφος αφορά τα άτομα τα οποία θα εκλεγούν, η δεύτερη αφορά τα κόμματα. Και η κλίδα της κατανομής των εδρών στο Κοινοβούλιο δεν τροποποιείται, αλλά υπάρχει η δυνατότητα να επιλέγονται διαφορετικά οι υποψήφοι συγκεκριμένοι. Επομένως, αυτή είναι λοιπόν μια λύση η οποία μπορεί να ξεπεράσει τις αντιρρήσεις και των δύο πλευρών και θα κάνει πιο δυνατή την έγκριση και στην Ολομέλεια. Τέλος, θέλω να υπενθυμίσω ότι οι συνάδελφοι οι οποίοι είχαν εκφράσει αμφιβολίες και αντιρρήσεις ε, έχουν δει τις αντιρρήσεις αυτές να καλύπτονται από τον Άντριου Νταφ, θα έπρεπε αυτοί οι συνάδελφοι να έχουν το θάρρος να υποστηρίξουν αυτή την πρόταση στην Ολομέλεια, γιατί με τον τρόπο αυτό νομίζω θα μπορέσουμε να κάνουμε όλοι ένα βήμα προς τα εμπρός. Ακόμη τρει τοποθετήσει Πήγε 12.30 και πρέπει οπωσδήποτε να τελειώνουμε. Παρακαλώ να είστε πολύ σύντομοι. Kiitoksia, herra Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να δείξω δύο θέματα. Καταρχάς, νομίζω ότι ξέρετε ότι ο κόσμος Ασφαλώς και έχει όνειρα, έχει φιλοδοξίες και η ζωή σημαίνει ότι δεν ξέρουμε τι θα φέρουν τα όνειρά μας πάντα. Σήμερα συζητάμε 50 διαφορετικά όνειρα τα οποία μπορούμε και προσπαθούμε να συνενώσουμε σε ένα. Κάποια μπορεί να είναι πολύ σημαντικά. Θα πρέπει να δεχτούμε όμως ότι υπάρχουν και καινούργια όνειρα, καινούργιοι στόχοι, οι οποίοι ίσως να είναι και καλύτεροι. Για να έρθω τώρα στα δύο σημεία που ήθελα να αναφέρω. Καταρχάς, για το κοινό ευρωπαϊκό κατάλογο και ψηφοδέλτιο αναφέρθηκε προηγουμένως και σας το έχω πει και στο παρελθόν ότι εμένα δεν με ενθουσιάζει η ιδέα. Και παρακολουθώντας και την όλη συζήτηση πρέπει να σας πω ότι όλο και λιγότερο ενθουσιάζομαι. Γιατί φαίνεται ότι υπάρχουν καλοί και κακοί πανευρωπαϊκοί βουλευτές. Έχουμε λοιπόν τους 25 καλούς Ευρωπαίους ε, στον συνολικό κατάλογο, στον πανευρωπαϊκό κατάλογο και οι υπόλοιποι δεν είναι καλοί. Τι να σας πω, εγώ πραγματικά δεν το υποστηρίζω αυτό ως προσέγγιση. Εγώ είμαι εκλέχθηκα. Αν είχα εκλεχθεί από τον κατάλογο αυτό, σας ρωτώ, τι ευθύνη δεν θα είχα απέναντι στους εκλογείς μου. Εγώ θεωρώ ότι η δημοκρατία συνεπάγεται και κάποιο είδους δέσμευση. Αν η Φιλανδία, λοιπόν, αποτελεί μία ονιαία εκλογική περιφέρεια, αυτό για μένα είναι προβληματικό, γιατί θα πρέπει να ταξιδεύω δηλαδή σε όλη τη Φιλανδία. Αυτό θεωρώ ότι παρουσιάζει προβλήματα. Και επίσης μήπως το Κοινοβούλιο θα πρέπει να αποφασίσει κατά πόσο το προσθεθούν επιπλέον ή όχι αυτοί οι... Συγγνώμη κυρία Τερμέκη, πέντε λεπτά μας μείνανε και πρέπει να μιλήσουν και άλλοι δυο. Λοιπόν, και μετά πρέπει να απαντήσει και ο κύριος Νταφ. Παρακαλώ να είστε πάρα πολύ σύντομοι tämä vienti tänne neuvoston kokoukseen. Ναι. Τέθηκε το θέμα της διάσκεψης του Συμβουλίου. Νομίζω ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να αποφασίσει πρώτα επί της απόψής του και μετά να προβεί σε διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Και αυτό αφορά μόνο μία μικρή, ένα μικρό τμήμα των Ευρωβουλευτών. Νομίζω ότι η δημοκρατία θα πρέπει να έχει πιο ευρία βάση. Ο κύριος Γουαλτιέρη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εγώ πιστεύω ότι όλα αυτά που συμβαίνουν με την κρίση και τα προβλήματα, τα οικονομικά και δημοσιονομικά προβλήματα ε, αποδεικνύουν ότι η Ευρώπη είναι απαραίτητη. Χωρίς Ευρώπη δεν μπορούμε να διακυβερνήσουμε οικονομικά. Πριν από τα τέλη της θητείας, δεύτερον αυτό, ξέρετε ότι θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τις διάφορες κοινοβουλευτικές έδρες εν ώψη της εισόδου νέων μελών. Πρέπει να αντιμετωπίσει λοιπόν το κοινοβούλιο αυτό το πρόβλημα. Η σοσιαλιστική και δημοκρατική ομάδα υπερψήφισε την έκθεση DAF σε αυτή την επιτροπή και δεν θα είχε κανένα πρόβλημα να κάνει το ίδιο στην Ολομέλεια. Φυσικά καταλαβαίνω ότι είναι αναγκαίο να έχουμε μια ευρεία συνένεση. Οπότε και εμείς συμφωνήσαμε με την ιδέα του να επανέλθει η έκθεση στην Επιτροπή. Καταλαβαίνουμε επίσης και την πολυπλοκότητα μιας τροποποίησης της συνθήκης. Υποστηρίξαμε κατά συνέπεια και όλη αυτήν την ε, ε, λογική, ε, τη γραμμή ευελιξίας, δηλαδή την θέση Höfner για μια υπερεθνική λίστα, για ένα υπερεθνικό ψηφοδέλτιο. Ο εισηγητής θέλει να ξεκινήσει έναν διάλογο με το Συμβούλιο και να ξεκινήσει διαπραγμάτευση πριν από την έγκριση της έκθεσης υπάρχει προηγούμενη συνένεση η διαπραγμάτευση για τις εξωτερικές ε, υπηρεσίες της Ένωσης ε, <coughs> ψηφίστηκε στην Επιτροπή και μετά επικύρωσε την ψηφοφορία η Ολομέλεια. Πρόκειται για μια διαδικασία η οποία δεν εντάσσεται στη παραδοσιακή διαδικασία της συναπόφασης. Εμείς δεν έχουμε αντιρρήσεις σε αυτή τη διαδικασία. Πρέπει όμως να ξεκαθαρίσουμε επί ποιας βάσης θα διαπραγματευτούμε. Είτε επί της βάσης αυτών που έχει ήδη ψηφίσει η Επιτροπή μας, δηλαδή την παλιά έκθεση DAF, είτε βάσει αυτού του νέου κειμένου το οποίο θα πρέπει να ψηφίσουμε. Υπάρχει, επειδή είναι και του ιδίου συντάκτη, υπάρχει σαφώς ε, συμβατότητα μεταξύ των δύο κειμένων. Εμείς ε, πάντως ε, θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε βάσει της θέσης της Επιτροπής μας μια διαπραγμάτευση με το Συμβούλιο. Εγώ έχω τον Μπρος και πραγματικά παρακαλώ δηλαδή. Και εγώ τον αντίον της παραγράφου 2 σε σχέση με την λίστα των 25 πανευρωπαϊκών βουλευτών. Η δημοκρατία σημαίνει κυβερνήση από, τους λα... από το λαό με μία ε, ενιαία ταυτότητα και ένα ενιαίο χώρο. Δεν είναι η κυβέρνηση από ένα αυθαίρετο αριθμό ατόμων. Μπορεί να περιμένει ο κ. Δάφο ότι κάπου θα υπάρξει πανευρωπαϊκή ταυτότητα, αλλά υπάρχουν πολλοί που έχουν διαφορετική γνώμη. Αυτή τη στιγμή όμω είναι σίγουρο ότι δεν υπάρχει. Μια πανευρωπαϊκή εκλογή με πανευρωπαϊκά κόμματα χωρί μια προηγούμενη κοινή ταυτότητα θα είναι ούτω ή άλλω ακατανόητη για πολλού εκλογή και θα υποστηρίξει περισσότερα τα κόμματα τα οποία θέλουν μια πανευρωπαϊκή προσέγγιση και θα είναι εναντίον των κομμάτων που δεν θέλουν μια τέτοια προσέγγιση. Ευχαριστώ κύριε Ντάφε για την απάντηση. Αλλά τώρα επειδή τελειώνουμε το χρόνο να προτείνω το εξή. Ε, αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Η συνθήκη της Λισαβόνας προβλέπει έναν ενιαίο εκλογικό νόμο. Οπότε η ιδέα του να κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να μην μας απορρίψουν και δεύτερη φορά στην Ολομέλεια μου φαίνεται απόλυτο λογικό. Φυσικά και μου φαίνεται λογικό μια ασθενή ένας, ε, ε, μια ομάδα βουλευτών να διαπραγματευτεί με το Συμβούλιο. Αλλά δεν μπορούμε όμως και να απογυμνώσουμε αυτή την Επιτροπή από τις εξουσίες της. Φυσικά και θα πρέπει κάτι να γίνει, να ψηφίσουμε. Λοιπόν, Νταφ, αυτό το διαδικαστικό δεν μπορούμε να το δούμε την επόμενη εβδομάδα στη συνεδρία των συντονιστών. Ναι, κύριε Πρόεδρε, θα μπορούσαμε. Δεν είμαι σίγουρος τι θα κερδίζαμε με τον τρόπο αυτό. Εκτιμώ όλα αυτά τα σχόλια. Θα έλεγα στον κύριο Φόξα εδώ ότι με ζήτησε η Επιτροπή μας να παραμείνω πιστός στο βαθμό του δυνατού στις αρχές που είχαμε θεσπίσει στην πρώτη έκθεση. και δεν θα αποστραφούμε από αυτούς τους στόχους όταν πλησιάζουμε το τέλος της διαδικασίας. Ήταν σε μία μειοψηφία ο κύριος Φόξ και ο κύριος Πρόντς αλλά οι περισσότεροι βουλευτές στην Επιτροπή μας υποστήριξαν την ιδέα μιας πανευρωπαϊκής λίστας. Θα έλεγα στον κύριο Μπρόνς, δεν υποστηρίζω μια πανευρωπαϊκή ταυτότητα, αν υπάρχει κάτι τέτοιο. Υποστηρίζω όμως μια μεταεθνική ταυτότητα. Και κάτι τέτοιο νομίζω το δέχονται πάρα πολλοί πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το οποίο θα ήθελα σαν διαδικασία να θεσπίσουμε είναι να υπάρξει μια προθεσμία για τροπολογίες και να ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας, να συζητήσουμε, να συνεχίσουμε τη συζήτηση για το τι θα συμβεί στη συνέχεια, αν θα ζητήσουμε από την συνέλευση των Προέδρων για να συζητήσουμε άτυπα με το Συμβούλιο ή όχι. γιατί χρειαζόμαστε την υποστήριξη του Συμβουλίου και της Επιτροπής για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε ένα φάκελο όπως αυτόν, ένα θέμα όπως αυτό. Και νομίζω ότι αυτό είναι λογικό και σκόπιμο και χαίρομαι που ο κύριος Κουατιέρη και ο κύριος Έφνερ συμφωνούν μαζί μου στο σημείο αυτό. Ο κύριος Σόπλη ζήτησε μία περίοδο περισυλλογής. Μάλιστα, αλλά θα πρέπει να είναι πολύ τολμηρή η περισυλλογή αυτή. Ιδάλλως, η νομιμότητα και αν θέλετε η μειούμενη δημοτικότητα του Κοινοβουλίου κυβεύεται περιπτέρω. Πρόεδρε, λοιπόν, με όλο το σεβασμό θα ήθελα να θέσουμε μία προθεσμία καταληκτική για την κατάθεση των τροπολογιών. Η γραμματεία μου προτείνει 26 Οκτωβρίου. είναι Una sufficiente riflessione. Può andare? Σύμφωνοι. Ούτως ε, συμφωνείτε. 10 Οκτωβρίου από τις 3 μέχρι τις 6.30 την ε, Τρίτη το πρωί από τις 9 ως τις 12.30. Πέρας τη συνεδρίαση. Θυμάμαι κάθε φορά ότι είμαι δικαστής και αντί να λέω πέρας τη συνεδρίαση, λέω πέρας τη συνεδρία.